Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ, καθίστε για να συνεχίσουμε. Όπως συμφωνήσαμε και χθες, θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Μωράν Σερτιέ που θα μας ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, Χθε ξεκίνησε ο ένατος τριμερής διάλογος με μια ερώτηση που θέσαμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αντίκτυπο των αποφάσεων και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εγώ προσωπικά, αλλά δεν ήμουν η μόνη που είχα αυτή την αίσθηση, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι σε πολλές πολιτικές ομάδες την ίδια εντύπωση αποκόμισαν, ότι οι αναγγελίες που έγιναν γιατί τη σχέση του Ταμείου Βοήθειας στους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, δεν εξασφαλίζονται. Και σίγουρα οι προϋποθέσεις πρόσβασης στα δύο ταμεία είναι διαφορετικές. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, χθες ε, το βράδυ συζητήσαμε εκτενώς για το ποιο, ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Ταμείου αυτού και μάλιστα είχαμε και σφοδρές συζητήσεις για το θέμα αυτό, γιατί αφενός τα επιχειρήματα του Συμβουλίου μένουν αμετάβλητα. Πρώτον, δεν υπάρχει νομική βάση. Δεύτερον, αυτό, οι δικαιούχοι δεν ε, είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Και όλο το βράδυ το Συμβούλιο προσπαθούσε να μας αποδείξει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης αφορούσαν ε, το κοινό στόχο, το, το, το κοινό που είναι ο στόχος, Δικαιούχου ε, δικαιούχους, αποδέκτες του Ταμείου, κάτι που δεν ε, ήταν αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Στις διαπραγματεύσεις ε, μας παρέχει ανεκτήμητη βοήθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ το Συμβούλιο θεωρώ ότι στηρίζεται υπερβολικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που χθε δεν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το άρθρο 3, κάποια πρόοδο παρόλα αυτά σημειώθηκε. Και πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις μας και ο τρόπος που άσκησα εγώ τις διαπραγματεύσεις δεν εκτράπησαν από το πλαίσιο που θέσαμε με τη διαπραγματευτική εντολή. Γιατί η διαπραγματευτική μας εντολή ήταν σαφέστατη και προέκυψε από συγκεκριμένες πλειοψηφίες και αυτή τη γραμμή ακολουθούμε απερίσπαστη απέναντι στο Συμβούλιο. Αυτά κυρίες και κύριοι, με δύο λόγια, για τις χθεσινές διαπραγματεύσεις. Και σίγουρα άλλο τρόπο διαπραγμάτευση χρησιμοποιούμε τώρα στην Ελλανδική Προεδρία από αυτό που είχαμε στην Κυπριακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευκολότερες οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο, υπάρχουν απορίες, ε, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Να προσθέσω σε σχέση με αυτά που σωστά μας είπε η συγγήτρια, ότι όπως και για άλλα θέματα, για μας το βασικό διακύβευμα των διαπραγματεύσεων είναι να εξακριβώσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα συμπεράσματα της 8 Φεβρουαρίου θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Γιατί πέρα το Ταμείο για τη βοήθεια στους απόρους, είχαμε το, τα 3 3 δισεκατομμύρια για, το, για την εγγύηση για τους νέους, που συνδέονται πια με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κάτι που προϋποθέτει αλλαγή των νομικών βάσεων. όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και για τη Γενική Νομοθεσία. Τον κανονισμό, δηλαδή, των κοινών διατάξεων, Common Provision Regulation, και γι' αυτό έχουμε δύο μεθόδους πιθανές. στο, στο τέλος του τριμερής διαλόγου θα μας υποβάλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα πρέπει να δούμε πώς θα θετήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ε, τρο... τροποποιήσεις, δηλαδή μια αναθεωρημένη έκδοχη. Δύο εβδομάδες και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, υποβάλει προτάσεις. Μάλλον θα υπήρξαν εντάσεις και τριβές με το Συμβούλιο. Βέβαια η Ιρλανδική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί αν ε, δεν λάβει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο φοβάται το νομικό κενό και θα αναλάβει πρωτοβουλία η Ιρλανδική Προεδρία. Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και μάλιστα πάρα αυτά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το έργο της. Αλλά Κάποιες προτάσεις κατευθυντήρες για θα πρέπει να υπάρχουν για την τροποποίηση των νομικών βάσεων. Δεύτερο σχόλιο για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων ως προς το CPR. Common Regulation Provision. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι σε κάποιες ομάδες Εργασία του Συμβουλίου ακούστηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί ή να παραιτηθεί το 25% υπέρ του ΙΕΦΣ και 20% υπέρ του στόχου της ένδυας. Δεν είναι αυτή όμως η κρατούσα γνώμη στην Επιτροπή Απασχόλησης, στη δική μας. Εξού και η ανάγκη όσων είστε μέλη και στις δύο επιτροπές να επιμείνετε και στις δικές μας προτεραιότητες ώστε να περάσει το μήνυμά μας και μέσω του εισηγητού μας, του κυρίου Άνταμ Κόζα για τη σημασία που αποδίδουμε στο θέμα αυτό που αφορά το άρθρο 84 του κανονισμού για την οποία υπάρχει κοινή αρμοδιότητα πολλών επιτροπών. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο, οπότε κυρία Μωράν Σαρτιέ, για να ολοκληρώσει. Θα ήθελα να στενιστώ και εγώ την ανάλυση σας και να διευκρινίσω ότι χθες το βράδυ στις συζητήσεις, για να μην πω στις μάχες που είχαμε με το Συμβούλιο για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Ταμείου, διαπιστώσαμε ότι το Συμβούλιο επέμεινε στο θέμα του κατά πόσο θα αφήσουμε 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους απόρους, ε, τους αναξιοπαθείς, για να τους βοηθήσουμε να καταπολεμήσουν την ένδια. Αυτό το θέμα βρέθηκε στην καρδιά των συζητήσεων και αποτέλεσε βασικό επιχείρημα του Συμβουλίου. Χρειάστηκε να αναπτύξουμε όλα μας τα επιχειρήματα με επαναφορά στο θέμα αυτών των δικαιούχων και του στόχου της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τελειώσαμε λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα στην μέση διάταξη. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 20, 23, συγγνώμη, λέει πρόεδρος, 23. Κοινωνική κατοικία λοιπόν, η κοινωνική στέγαση. Η κυρία Ντελή Χαίρομαι που σας παρουσιάζω σήμερα την πρώτη διατύπωση, την πρόταση της έκθεσής μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεισήγητες και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και στο στάδιο της τροπολόγησης. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσες αρμοδιότητες στον τομέα της κατοικίας και της κοινωνικής κατοικίας. Έμεσα όμως εμπλέκεται. Ε, επιδοτήσεις, κοινωνική σύνοχη, ανάπτυξη της υπαίθρου, ενεργειακή αποδοτικότητα, δημοσιογραφικές ε, αλλαγές. Γενικά βλέπουμε ότι έχει στη διάθεσή της ε, πολλούς μοχλούς δράσεις και έμεσα και άμεσα μέσω της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική αυτή πρωτοβουλίας λοιπόν είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν οι λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 25 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών κατοικούν σε ε, κτίσματα που ε, ανήκουν στην κοινωνική κατοικία. Όλες οι χώρες έχουν τέτοιες κατοικίες εκτός από την Ελλάδα βέβαια ποικίλουν ε, τα ποσοστά ανάλογα με χώρες, ανάλογα με τις περιφέρειες, τις αστικές περιοχές, στο κέντρο των αστικών περιοχών, στην περιφέρειά τους. Βασικός μου στόχος είναι να επιβεβαιώσουμε ότι το δικαίωμα στην κατοικία είναι θεμελιώδες δικαίωμα που καθορίζει το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή και θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να το θέσουν σε εφαρμογή. Με την κρίση δυστυχώς ε, ταλανίζεται το συγκεκριμένο δικαίωμα και γίνονται πολύ δύσκολες οι δυνατότητες πρόσβασης στην κοινωνική κατοικία λόγω και της αύξησης των ενοικίων και του κόστους ενέργειας. Το 2010 σχεδόν 5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υπέφερε σε επίπεδο κατοικίας, ενώ το φαινόμενο αυτό των ε, αστέγων ουσιαστικά συμπολιτών μας δεν θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα. Ένα 14% ζούσε σε κατοικίες απαράδεκτες και 10,4% πλήρωνε πάνω του 40% του εισοδήματός τους για ενίκιο ή για την κτήση της κατοικίας που κατήχαν. Λοιπόν, πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία έχει δημιουργήσει η οικονομία της αγοράς στο επίπεδο της κατοικίας και να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα σε μια κατοικία αξιοπρεπή με προσβάσιμη και εφικτή για όλους δυνατότητα ε, κατοίκησης. Δυστυχώς ε, οι περικοπές οι δημοσιονομικές μειώνουν τις δυνατότητες αυτές και φυσικά η ιδιωτική αγορά από μόνη της δεν καλύπτει τις ανάγκες πρωτοβουλία λοιπόν, η έκθεση πρωτοβουλίας μάλιστα είναι να προωθήσει ακριβώς την κοινωνική κατοικία για να βγούμε και από την κρίση. Γιατί πρώτον θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο και τη σημασία των επενδύσεων στον τομέα. Ο ΙΕ και ο ΑΣΑ έχουν περισσότερες, ε, ε, περισσότερα στοιχεία και περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους για την κοινωνική κατοικία. Απαιτείται ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκό με βάση συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για να καταπολεμήσουμε την μάστιγα και της αδυναμίας πρόσβασης στην ενέργεια και γενικά θα είναι κάτι το χρήσιμο. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με τα θέματα της κατοικίας σαν έναν από τους παράγοντες πτώχευσης ουσιαστικά ε, των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Πρέπει λοιπόν οι επενδύσεις στην κοινωνική κατοικία να θεωρηθούν σαν πιο σημαντικές στα πλαίσια της οικονομικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Είναι στρατηγική η σημασία τους στα πλαίσια ενός συμφώνου κοινωνικών επενδύσεων. Θα πρέπει επίσης ο ρόλος του μακροοικονομικού σταθεροποιητή του τομέα αυτού να γίνει αντικείμενο καλύτερης αναγνώρισης με αύξηση των κοινωνικών κατοικιών. Έτσι θα αποφύγουμε ε, τις φούσκες στον τομέα της αγοράς κατοικίας. Δυστυχώς αυτού του είδους οι καταστάσεις έχουν παίξει τραγικό ρόλο τελευταία. Βλέπουμε τι συνέβη στην Ισπανία με την κατοικία. Καλύτερα λοιπόν να προλαμβάνει κανείς και να προσφεύγει με αυξημένο ρυθμό στην χρήση αυτού του μοχλού που είναι η κοινωνική κατοικία. Χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας λέγοντας ε, ακριβώς και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020. Θα πρέπει λοιπόν έτσι να προχωρήσουμε και προς την ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση για την αηφορία και τον διεθνή ανταγωνισμό. Γι' αυτό τα ταμεία της συνοχής θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο είτε υπέρ της πρόσβασης σε ενεργειακές υπηρεσίες ποιότητας από ανανεώσιμες πηγές και στην κάλυψη των αναγκών ευάλωτων κοινωνικών πληθυσμών όπως η Ρωμά και οι Άστεγοι, ανταποκρινόμενοι στις δημοκρατικές αλλαγές. Το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο θα επιτρέψει την χρηματοδότηση των προσπαθειών κατάρτισης και στον τομέα των νέων θέσεων απασχόλησης στον πράσινο αν θέλετε ορίζοντα. Στα πλαίσια λοιπόν της στρατηγικής 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δανειοδοτικές δυνατότητες και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί το μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ στον τομέα της των κατασκευών και της οικοδομής. Έτσι θα ανταποκριθούμε στην κατεπίγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, και έτσι θα δώσουμε εγγυήσει και στην κατανομή των κατοικιών για να μην υπάρχουν διακρίσεις και να μην υπάρχουν προσπάθειες αποφυγής των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Εδώ το θέμα της διαχείρισης της κοινωνικής κατοικίας τίθεται. Τίθεται επίσης το θέμα της δυσκολίας πρόσβασης στην ενέργεια. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ορίσουν σωστά το φαινόμενο αυτό το οποίο αφορά σήμερα 50 με 55 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Θα πρέπει από τη μία να υποστηρίξουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλέον ενεργοβόρων κατοικιών μέσω χρηματοδοτικών μέσων αποτελεσματικών μέσω πρόθεσμα και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε, να θέσουμε την δυνατότητα μέτρων ελάφρυνσης των, του κόστους της θέρμανσης για τις κατοικίες. Ελπίζω λοιπόν η έκθεση αυτή να είναι ένα μήνυμα για το σύνολο αυτών που ζουν σε κακές κατοικίες στην Ευρώπη και φυσικά υπέρ των αστέγων και εύχομαι να το υποστηρίξετε και να συνεισφέρετε και εσείς με τον δικό σας τρόπο. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Μπερές. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα δώσω σε κάθε έναν που θα πάρει το λόγο δύο λεπτά. Πρώτα ο κύριος Σόγκορ και μετά ο κύριος Σέρκας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο την κυρία Νταλή για την πρωτοβουλία διοργανώσαμε και ακροάσεις και νομίζω ότι καταφέραμε να λάβουμε πληροφορίες εις βάθος για το συγκεκριμένο τομέα. Πρόκειται για ένα πολύ επίκαιρο θέμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό για να το συζητήσουμε σε τέτοιου καιρού κρίση. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή και στέγαση με υγιεινούς όρους ε, στέγασης, γιατί χιλιάδες άτομα χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις στατιστικές του της ΠΟΗ για την στέγαση, για την χρηματοδότηση που αναφέρει ότι ο κόσμος πολύ συχνά πληρώνει 55% των εισοδημάτων του για την στέγαση ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό αυτό. Επίσης μιλάει ε, σε ό,τι φορά το προσδόκιμο ζωής η έκθεση για την επιρροή της στέγασης. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα και έχει αποδεχτεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μόνωση, για παράδειγμα, του σπιτιού. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής. Ε, θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες σε ό,τι αφορά την στέγαση κυρίως για τους νέους, για τους πρεσβύτερους και θα τονίσω ιδιαίτερα τα θέματα διαφοράς γενεών σε ό,τι αφορά τα θέματα στέγασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σέρκας και μετά ο κύριος Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι από τα πιο σημαντικά θέματα της κοινοβουλευτική μας θητείας, γιατί θεωρούμε ότι η στέγαση στο δικαίωμα στην κατοικία μαζί με το δικαίωμα στην απασχόληση και η έλλειψη για το δύο είναι από τους χειρότερους εχθρούς ε, του ανθρώπου που δεν μπορεί έτσι να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπέ σχέδιο για το βιωτικό του επίπεδο και τη ζωή του. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πάνω από 150 εκατομμύρια Ευρωπαίους με προβλήματα κατοικίας και 2 εκατομμύρια των συμπολιτών μας δεν έχουν καν σπίτι. Το πρόβλημα είναι σοβαρότατο και ξεπερνάει την κρίση. Αποτελεί την, έκφραση, την έκφανση ενός διαρθρωτικού προβλήματος ή την έλλειψη δημόσιων πολιτικών στέγασης. Και υπάρχει απόλυτη αδιαφορία μερικές φορές σε κοινωτικό επίπεδο για το θέμα αυτό. Γι' αυτό είναι και πολύ εύστοχη έκθεση. Και ευτυχώς η κυρία Καρή Μαντελή περιλαμβάνει στην έκθεσή της όλες μας τις ανησυχίες. Γι' αυτό και θα είναι πολύ εύκολη και απρόσκοπτη η συνεργασία μας. Επίσης να υπογραμμίσω ότι ίσως θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη σειρά των προτεραιοτήτων για να είναι πιο εμφανές το μήνυμά μας. Πρώτα να αναλύσουμε τα προβλήματα, ε, τις αιτίε τους, τις ρίζες τους και μετά να προτείνουμε λύσεις για να είναι πιο ευανάγνωστη από πολιτική άποψη η έκθεση και το, κείμενο της έκθεσης. Αυτό προσπάθησε να κάνει και η Καρή Μαντελή, αλλά χρειάζεται μια καλύτερη ανακατάταξη των σημείων για να είναι πιο ευανάγνωστο το κείμενο. Για μας τους σοσιαλιστές είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να το επιλύσουμε βέβαια με μέτρα, αλλά και να το προλάβουμε. Γιατί δεν αρκούν ε, οι θεραπείες, ε, δεν αρκεί η ίαση, χρειάζεται και η πρόληψη, να αποφύγουμε την δημιουργία των προβλημάτων, γιατί μερικές φορές είναι και θέμα πρόληψης αυτή η πολιτική στέγασης. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση, να μην περιοριζόμαστε από το στενό εθνικό πρίσμα. Και φυσικά αυτό το θέμα θα συνδυαστεί με τη συζήτηση για, την, ε, για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ και το θέμα της ανταγωνιστικότητας που πλήττει πολλές εθνικές πολιτικές. Ο Φιλ Μπενιό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία τη σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται ε, και εμπλέκει τους σκιώδεις ε, εξ αρχής την ε, δουλειά της. Και σε ό,τι αφορά και τις ακροάσεις, να την ευχαριστήσω που συμπεριέλαβε κάποιες από τις ιδέες που και εγώ τις υπέβαλα σε αυτή τη φάση του σχεδίου. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο τι έγινε με την πρόταση δημιουργίας μιας νέας υπηρεσίας πού θα εντασσόταν αυτή η υπηρεσία και με, σε ποια, με ποια χρηματοδότηση. Γιατί προφανώς στα πλαίσια του σε δημοσιονομικού πλαισίου και των σχετικών διαπραγματεύσεων θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, θα επηρεάσει αυτό τον ε, προπολογισμό με το ESF και κατά πόσον έχει σκεφτεί και άλλους μηχανισμούς ε, για την επίτευξη των ίδιων στόχων, ίσως μέσω υφιστάμενων υπηρεσιών. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, σε μεγάλο βαθμό θα είναι διευκρινιστική φύσεως και θα προσθέσουν και κάποια στοιχεία. Θα ήθελα να τονίσουμε το, την πτυχή της ενεργειακής αποδοτικότητας και το κατά πόσο μπορούμε μέσω καινοτομικά συστήματα, μέσω μόνωσης, μέσω φτηνών σπιτιών ε, να βοηθήσουμε τους ε, ιδιαίτερα ευάλωτους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Έχουμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα που εντάσσεται στο Green Deal και εφαρμόζεται από την κυβέρνησή μα και θα ήθελα κάποιε από τι προτάσει αυτέ που έχουν συμπεριληφθεί να τι καταθέσω ω τροπολογίε. Ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε υπερβεί κάποιε αρμοδιότητέ μα. Η συγκίτρια, ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι ήταν πολύ περιοριστική και αυστηρή προκειμένου να μείνουμε στον τομέα των αρμοδιοτήτων μας. Ε, υπάρχουν κάποιοι τομείς που θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και προσβλέπω σε μετέπειτα στην συνεχιζόμενη συνεργασία με την εισηγήτρια της επόμενης εβδομάδας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πώς θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Μάλιστα. Τότε να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Ντελή. Ευχαριστώ. σημείωσα προσεκτικά και θα λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις των συνεισηγητών. Και στην επόμενη συνεδρία σας εξηγήσω γιατί είναι απαραίτητη η σύσταση αυτού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Στέγασης η κατοικίας. Γιατί αυτή τη στιγμή στερούμαστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οποιασδήποτε στρατηγικής ώστε να περάσουμε από τις θερτικές των αστίγων για τις κακή στέγασης, να περάσουμε από την, ε, την επισφαλή κατάσταση της ενέργειας ε, ε, στο θέμα της διακυβέρνησης. Όλοι αυτοί οι δείκτες που είναι σημαντικοί δεν είναι στη διάθεσή μας σήμερα. Οπότε καμία χώρα δεν καταφέρνει να επιλύσει την κρίση στη στέγαση, να προλάβει τις φούσκες των ακινήτων ή την εκτείναξη στα ύψη των τιμών ακινήτων. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο παρατηρητήριο. Γι' αυτό και μα είναι απαραίτητο για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα, για να επικεντρωθούμε και στην πρόληψη και όχι μόνο στη θεραπεία. Και σίγουρα έχετε δίκιο ότι το δικαίωμα στην κατοικία είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Και θα πρέπει όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν δικαίωμα σε αυτό και πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα. Αυτά και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου ξαναδώσατε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Να προσθέσω εδώ ότι στα πλαίσια της διαδικασίας τροπολογιών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια της εξέτασης της συγκεκριμένης έκθεσης κάποιες συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει στα πλαίσια της εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, και στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα του. Μία από τις προτάσεις η οποία έχει πολύ συζητηθεί είναι η ένταξη των λεγόμενων κοινωνικών δικτών στον οδικό χάρτη που θα εξετάσει τις εξελίξεις ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ένας δείκτης που να αφορά την κοινωνική κατοικία είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται αντικείμενο συχνής αναφοράς. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνεχίσουμε με την πρόταση αυτή. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 20 7 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι. Λίγη ησυχία παρακαλώ λέει η Πρόεδρος. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της 20 Μαρτίου και θα τις αναλύσουμε στις 22 Απριλίου για να περάσουμε στις 23 σε ψηφοφορία έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την Ολομέλεια του Ιουνίου. Φτάνουμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία είναι στο σημείο 24 το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την οδηγία 2009-13 από πλευράς Συμβουλίου και της Συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις μεταφορές για να διευκρινηθεί η εντολή από πλευρά Συμβουλίου και να διασφαλιστεί η νομική συμβατότητα των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, αποφασίσαμε να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια οι τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης όπως και αυτές που προβλέπονται στην σύμβαση, ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Εμπορική Ναυτιλία. Αυτά μπορούν να προστεθούν στη νομική βάση που θα χρησιμοποιηθεί για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια λοιπόν θα γίνει επί των τροπολογιών, όχι όμως επί του νομοθετικού ψηφίσματος μόνο και μόνο για να ξεκινήσει η συζήτηση με το Συμβούλιο. Θα εκφραστούμε λοιπόν επί της αρχής έτσι ώστε να ψηφίσει η Ολομέλεια τον τρόπο ορισμού της διαπραγματευτικής εντολής. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας επί της αρχής παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Yeah. Cette procédure est donc Η διαδικασία αυτή λοιπόν γίνεται δεκτή με τέσσερις ψήφους κατά. Κοιτάξτε, αφήστε με να ανακοινώσω το, την κατάληξη της ψηφοφορίας. Αυτό το αίτημα επικύρωσης λοιπόν της εντολής από την Ολομέλεια γίνεται δεκτό. Τέσσερις ψήφισαν κατά, μηδέν αποχές, έχετε το λόγο χωρίς ε, μικρόφωνο ο μιλητής. Δεν έχω την κάρτα μου, ζητώ να ψηφίσω ε, διανατάσεως χειρός. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν πρέπει να μας διακόπτεται. Θα καταμετρήσω την ψήφο σας και από εκεί και πέρα θα μας λέτε ε, όταν χρειάζεται. Τελειώνουμε με το 24 εν περιπτώσει. Θα ξεκινήσει η διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι τροπολογίες για τις οποίες ζητάμε να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 25, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, κοιτάξτε παρακαλώ ποιος δεν έχει την κάρτα του. Je Κοιτάξτε, με έκλεψαν. Μου έκλεψαν το πορτοφόλι, δεν έχω καν την κάρτα και δεν είχα και χρόνο να περάσω από το γραφείο μου. Ξεκίνησα τη δουλειά σήμερα το πρωί στις 8 και θα τελειώσω το βράδυ δυστυχώς στις 10.30. Συνεπώς για σήμερα τίποτα. Λοιπόν, 25. Απαλλαγή 2011 Γενικός Προϋπολογισμός Τμήμα Επιτροπή. Επαναλαμβάνω απαλλαγή 2011 Γενικός Προϋπολογισμός Τμήμα 3 Επιτροπή. Στην παράγραφο 1 έχω την τροπολογία 1 τσάμπα όρη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά την παράγραφο 1 έχω την τροπολογία 2 του ιδίου. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. Μετά την παράγραφο 5 έχω την 3 του ιδίου. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. Μετά την 8 έχω την τροπολογία 4 του κυρίου Ορή με προφορική τροπολογία από τον ίδιο τον εισηγητή. Την εισηγήτρια μάλλον. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Συνεπώς ψηφίζουμε την τροποποιημένη 4. Υπέρ, κατά, άποχες δεκτή. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Η απαλλαγή δίδεται. Στο 26 έχουμε την απαλλαγή 2011 για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το λεγόμενο σεντεφόκ Στην παράγραφο 1 έχω προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, δεν υπάρχει αντίρρηση, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 3, τροπολογία 1 του ορί, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. απολογία 2. Θέρκας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 40 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Η γνωμοδότηση αυτή συνεπώς γίνεται αποδεκτή. Φτάνω τώρα στην απαλλαγή 2011 για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βελτίωσης Συνθήκων ε, Διαβίωσης και Εργασίας. Μετά την παράγραφο 1 έχω την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Δεν υπάρχει αντίρρηση ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 3 έχω την τροπολογία 1 χάρκιν ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της απαλλαγής. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. «41 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Η απαλλαγή αυτή γίνεται δεκτή. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 28 στην απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ασφάλειας και Υγεία ε, που έχει έδρα το Μπιλμπάο, το Μπιλμπάο, όχι τη Βαρκελόνη, έκανα λάθος λέει πρόεδρος. Παράγραφος 1, προφορική ορολογία της εισηγήτριας. Υπάρχει κάποιος που είναι κατά. Όχι. Την θέτω σε ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Στην παράγραφο 1. Τροπολογία 1. Τσάμπα όρη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά την παράγραφο 3. Τροπολογία 2. Σέρκας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά την παράγραφο 3. Τροπολογία 3. Χάρκιν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 4, θέρκας, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Το σύνολο τώρα του κειμένου ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή. Δίδεται η απαλλαγή. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 29 για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μετά την παράγραφο 1 έχω την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 23 κατά. Οπότε δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία. Μετά την παράγραφο 1 έχω μια δεύτερη τροπολογία, προφορική πάντα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά την παράγραφο 2. Έχω την τροπολογία 1 όρη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρολικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 24 υπέρ. 16 κατά. Είναι σαφές γίνεται δεκτή. Και πάντα με την παράγραφο 2 έχω την τροπολογία 2 θέρκας. Με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 2 έχω την τροπολογία 3 χάρκινγκ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Θέτω στην ψηφοφορία το σύνολο ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 41 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Η έκθεση απαλλαγή γίνεται δεκτή, δίδεται η απαλλαγή. Περνάμε στο σημείο 30. Τελευταία απαλλαγή για το 2011 αφορά τις επιδόσεις στην δημοσιονομική διαχείριση των οργανισμών. Δύο είναι οι τροπολογίε, η μία αφορά την παράγραφο 2 του Jean Lambert, της Jean Lambert και είναι υπέρ κατά δεκτή. Στην παράγραφο 3 η συγγήτρια υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Δόθηκε η απαλλαγή. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 41. Εφαρμογή της οδηγίας 2085 ε, για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Πρόκειται για την έκθεση της κυρίας Γιούτα Στάινρουκ για την ε, νομική επιτροπή. Παράγραφος 1, τροπολογία 1 της, Άρια ΑΙΑ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. 22 υπέρ, 18 κατά. Τρεις εποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 2 της ίδιας συγκεκριτρίας Ε, Συντακτής είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, παράγραφος 3 του Φιλ Μπένιον. Ζητά διαγραφή. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 3, ποιο είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. «22 ψήφισαν υπέρ, 21 κατά». Εγκρίνεται και δίκιο είχατε που ζητήσατε έλεγχο. Παράγραφος 3, τροπολογία 3 του Φιλμπενιών. Ποιος είναι υπέρ, ζητά διαγραφή. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, δεύτερη συμβαστική τροπολογία υπέρ. Μα διαγράψτε το άρθρο, αγαπητέ συνάδελφε. Θα... Πρέπει να ξέρει κανείς τι κάνει στη ζωή. Α, συγγνώμη τώρα. Άκυρο. Ε, πέντε. Ποιο είναι υπέρ. Δεύτερη συμβαστική τροπολογία. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφό 6. Συμβαστική τροπολογία σε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Συμβαστική τροπολογία δέλτα υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 8, ε, συμβαστική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 8, τροπολογία 10 του Τζαμπαόρη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 11. Έχει αποσυρθεί, οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία F. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 γιατί 14 έχει αποσυρθεί. Ε, συμβαστική τροπολογία G. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται Γκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11 έχουμε την τροπολογία 17 του κυρίου Τσαμπαόρη. Ζητά διαγραφή. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 17. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 15 ψήφισαν υπέρ, 28 κατά και μία αποχή. Με διαφορά απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 11, τροπολογία 18 του κυρίου με τη μεγεψηφοφορία ψηφοφορία κατά τμήματα, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, το ζητά μέχρι το contract, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές εγκρίνεται, και το υπόλοιπο κείμενο τώρα υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 12, τροπολογία 19 του Φιλ Μπένιον. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, παράγραφος 20 και 21, γιατί είναι ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την γνωμοδότηση κυρία Στάιμπρουκ και τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 41 ε, υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Συγγετρία. Και περνάμε στο σημείο 32 ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση τη συνάντια Χέρι, προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Γνωμοδότηση που θα δώσουμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Παράγραφος 3. 1α. Ναι. Έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, 26 Jean Λάμπερτ και 27 Στίβεν Hughes και Evelyn Ρενιέ. Ψηφίζουμε από κοινού τι τροπολογίες 26-27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Για το άρθρο 6, παράγραφο 1 1F, τροπολογία 28 του Όλε Λούτβιξον. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το F, τροπολογία 29 τη Άρη Εσαϊά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 6. Παράγραφος 1α νέα. Συμβαστική τροπολογία α. Ε, ψήφισαν κατά οι φιλελεύθεροι, απορρίφθηκε. Άρθρο 6, ε, ε, συμβαστική τροπολογία α, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 4, τροπολογία 31, εσάια, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 6, παράγραφος 5, τροπολογία 32 της κυρίας εσάια, ποιος είναι υπέρ, ζητά διαγραφή, ποιος είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται άρθρο 7, παράγραφος 3, 33, τροπολογία του είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται άρθρο 7, παράγραφος 4 και τροπολογία 34 της κυρίας Ισάια. Ζητά διαγραφή. Προσοχή λοιπόν, αν θέλετε να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία, μην ψηφίσετε την τροπολογία αυτή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία σε ποιος είναι υπέρ τεσσάρων πολιτικών ομάδων, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία σε. Άρθρο 7, μετά την παράγραφο 4, 38, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 9, παράγραφος 1, η 39 καταπίπτει και η 40 το ίδιο. Οπότε πάμε στο άρθρο 14. Όχι, συγγνώμη, λάθος λέει η πρόεδρος. Η τροπολογία 40 Τζιν Λάμπερτ είναι συμβατή, οπότε ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 40, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 14, παράγραφος 3, 41, Στίβεν Hughes και Regner. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Στίβεν Χιούς και Ευλίν Ρενιέ. Ποιος είναι υπέρ, ζητά διαγραφή τροπολογία αυτή. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 17. Τροπολογία 43. Όλε κρίστερ και Ρενιέ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Άρθρο 22, παραγραφός 2 Δέλτα. Τροπολογία 44, Σαρίε Άια. Ποιο είναι υπέρ, κατά, Αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 45 της ιδέας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 46 της κυρίας Εσάια. Ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 23.4, 47 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 48 Κρίστενσεν. Μακερενιέ, Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 28, 4β. Τροπολογία 49. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε δύο πανομοιώτες τροπολογίες, την 50 Εσάια και την 51 για Κονσάρι. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Κεφάλαιο 4, 3, τίτλος. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 33, 5. Τροπολογία 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 33, 6. Τροπολογία 54 της κυρίας Εσάια. Ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 33, 7. Τροπολογία 55 της κυρίας Εσάια και πάλι διαγραφίζεται. ζητά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Μάλλον απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε όμως καλύτερα ηλεκτρονικά. Τροπολογία 55 που ζητά διαγραφή το άρθρο 37, 33 παράγραφος 7. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 18 ψήφισαν υπέρ, 25 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν, σαφέστατα. Άρθρο 34. Άρθρο 34 για τον τίτλο 56 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 34-1. Τροπολογία 57. Σαρίες Σάια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35-1. Εισαγωγικό τμήμα. Τροπολογία 58. Ρενιέ Κρίστινσεν Στάινρουκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 35.1α. Τροπολογία 59. Τζιν Λάμπερτ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 35.1β. Συμβαστική τροπολογία ε. Από τρει ομάδε. Ε, Συγγνώμη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται η συμβαστική F. Άρθρο 35. 1β. Α. Νέο. Τροπολογία 63. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 35.2. Τροπολογία 64. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. 65 συγγνώμη. Είναι συμβατή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ. Εγκρίνεται. Άρθρο 35. Παράγραφος 2. Υποπαράγραφος 1. Νέα. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα. Από πέντε ομάδες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική Δέλτα. Τροπολογία 35. Παράγραφος 5. Συμβαστική τροπολογία ΔΑ από δύο ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται, οπότε ψηφίζουμε την 67 τροπολογία των Ρενιά Κρίστενσεν και Στάινρουκ. Α, συγγνώμη, καλύπτεται από την προηγούμενη συμβαστική τροπολογία που εγκρίναμε, την D. Τροπολογία 68. Σάρι Σάια. Ναι. Ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 35-11. 69. Ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 43. 1β. Νέο. Τροπολογία 71. Ευλήν 9 Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Άρθρο 77, παράγραφος 1, τροπολογία 72, καταπίπτει. Και περνάμε στο άρθρο 78, παράγραφος 2α 9 τροπολογία 74, Στίβεν Χιούς, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 79, παράγραφος 3β, τροπολογία 75, Σάρια Σάια, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 81 1 β τροπολογία 77 Ισάια ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 81 1 σε τροπολογία 78 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 81 1 σε α ναι. νέο 79 Ισάια ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται και αυτή. Άρθρο 81, παράγραφος 3. Τροπολογία 80 της κυρίας Ισάια. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 82 για τον τίτλο. Τροπολογία 82, Τζιν Λάμπερτ. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 82.1. Συμβαστική τροπολογία G. Από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο άρθρο 82 μετά την παράγραφο 1. Συμβαστική τροπολογία Κ από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 82, παράγραφος 1α νέο. Τροπολογία 98, Πολμέρφη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 82, μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 99, Steven Hughes. Ποιος είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, αυτή καταπίπτει. Το ίδιο και η 100 και 101. Οπότε φτάνουμε στην τροπολογία 102, Jean Lambert. Αποχή από την εισηγήτρια. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Το ίδιο για την 103. της κυρίας Μενοδόρα Κλειβέτη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 103. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 19 υπέρ 24 κατά, χωρίς αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104, Ρενιέ. Ποιος είναι και τριοδέτερη; Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 82. 105 καταπίπτει. Το ίδιο και 106, 6 και 107. Άρα περνάμε στην τροπολογία, συμβαστική τροπολογία H, από πέντε ομάδες, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται για το άρθρο 82. Παράγραφος 2. Τροπολογία 118. Όλε Λούντβιγκσον ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 119. Σαρία Σάια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Υπέρ πρώτα, υπέρ. Για την 119. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 19 ψήφισαν υπέρ, 15 κατά. 8 αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Για το 82.1 σε η τροπολογία 118, η δικιά μου, θα πρέπει να ψηφιστεί. Ακόμη και να έχει εγκριθεί η ΔΕΛΤΑ συμβαστική τροπολογία, με εξαίρεση μία φράση. Το shall be entitled to relevant training. Α, όντως, έχετε δίκιο κύριε Λάμπερτ. Τροπολογία 112 λοιπόν, επαναρχόμαστε. Θα ψηφίσουμε... Τροπολογία 112 για το άρθρο 82 παράγραφος 1σε. Τροπολογία 112, Τζιν Λάμπερτ. Επειδή υπερψηφίστηκε η συμβαστική τροπολογία Δέλτα, θα ψηφίσουμε την τροπολογία χωρίς το shall be entitled to relevant training. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μια και η συμβαστική τροπολογία Δέλτα εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 112 της κυρίας Λάμπερτ, χωρίς όμως τη φράση θα δικαιούται κατάλληλη κατάρτιση. Shall be entitled to relevant training. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται την τροπολογία 112 της κυρίας Λάμπερτ. Άρθρο 82.2, παράγραφος, ε, συγγνώμη, τροπολογία 120, Ουγγορεάνου. Είναι συμβατή με την 119. Ποιος είναι υπέρ της 120. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 120 του κυρίου Ουγγουρεάνου. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ψήφισαν 16 υπέρ, 23 κατά. Τέσσερις αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 122 λέει πρόεδρος, 120 ήταν. Μετά την παράγραφο 2 τώρα, τροπολογία 122 καταπίπτει και ψηφίζουμε την 123 Σάρια Σάια. Διαγραφή ζητά. ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία I από πέντε ομάδες. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 82, 3, μετά την παράγραφα 3, 128 τη συναντιαχείριση. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη 29α, 29α, η τροπολογία 11 καταπίπτει. Για την αιτιολογική σκέψη 34 ψηφίζουμε την τροπολογία 12 σε που ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται η 12, οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία Β υπέρ από 4 ομάδες. Κατά, Είστε κατά τη συμβαστική τροπολογία Β τώρα. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική τροπολογία Β. Κατά άποχες εγκρίνεται για το 75. Συμβαστική τροπολογία ε από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 123. Τροπολογία 19. Φιλίπ Ντεμπάκερ. Ποιος είναι υπέρ. κατά απόχες απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 124. Συμβαστική τροπολογία G από τέσσερις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά το 124, τροπολογία 25 της κυρία Νάντια Χίρς. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 3 κατά, 6 εποχέ. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Συγγετρία. Nous en venons Φτάνουμε τώρα στην ψηφοφορία επί της εκθέσεως ε, Τσάμπα Σόγκορ για την πρόταση κανονισμού για τις δημογραφικές στατιστικές. Έχουμε γνωμοδότηση από τις Επιτροπές ε, Γυναικών, την Νομική Επιτροπή. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, έχω την τροπολογία 28 της κυρίας Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 2. Παρα, άρθρο 2, παράγραφος 1. Η τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε θα ψηφίσουμε την 29 Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 29. Ψηφίζετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 υπέρ 15 κατά 0 αποχές σαφές ότι γίνεται δεκτό. Λοιπόν, έχω τώρα την τροπολογία 3. Σόγκορ και άλλων. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Κυρία Παπαλοπούλου, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31. Ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20 κατά, 7 αποχές δεκτό. Euh, τώρα, 32 και Μαρινέσκου. Ποιοι είναι υπέρ της 32, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέτουμε σε ψηφοφορία τώρα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στο εισαγωγικό κομμάτι τη συμβιβαστική α. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θέτουμε σε ψηφοφορία τώρα την τροπολογία 8 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τοπολογία 9 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ποιοι είναι υπέρ της 10. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τη συμβιβαστική β. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στο σημείο H, αγγλικό, έχω την 38 της κυρίας Παπαδοπούλου και την 7 της περιφερειακής. Είναι ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ των δύο, κατά, αποχές, δεκτές. Στο άρθρο 2, στο νέο H, έχω την 11 του εισηγητή, το οποίο δεν γίνεται παραδεκτό. Οπότε φτάνω στην 39 Κλειβέτη έχει αποσυρθεί η 39 και στο άρθρο 3 πλέον, παράγραφος 1, θέτω σε ψηφοφορία την 40 της κυρίας Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 41 καταπίπτει, 42 έχει αποσυρθεί ήδη. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 40. Άρχεται η ψηφοφορία για την 40. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ 19 κατά γίνεται δεκτή η 40 επαναλαμβάνω. Η 12 έχει καταπέσει. Ακόμα και η 3 της ΑΦΚΟ, όπως και η 8 της Ρέγγι. Φτάνω τώρα στο άρθρο 3. Έχω την 43 Σόγκορ. Ποιοι είναι υπέρ της 43 κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα φτάνω στην 44 Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 την 45 της κυρίας Παπαδοπούλου ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 καταπίπτει, το ίδιο και η 13, οπότε ψηφίζουμε τώρα την, στο άρθρο 3 παράγραφος 3 την 9 της Ρέγγι, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στην παράγραφο 4 θέτω σε ψηφοφορία την 10 της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων σε δύο τμήματα, ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, δεκτό, το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, α μικρό. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 γυναικών. που έχει καταθέσει το σύνολο της Επιτροπής και η κυρία Παπαδοπούλου. Η συγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1. Συμβιβαστική σε Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Φτάνουμε στο άρθρο 5 παράγραφος 1 νέο. Έχω την 55, έχει καταπέσει 55 και την 5 παράγραφος 1 ψηφίζουμε την 15. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Την 56 κυρίας Παπαδοπούλου ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 56 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας «26 υπέρ, 13 κατά, 3 αποχές» δεκτή. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 την 57 Παπαδοπούλου ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 5 παράγραφος 3 16 εισηγητής ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 της κ. Παπαδοπούλου ποιοι είναι υπέρ Συγγνώμη λέει η πρόεδρος λάθος. 58. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Ρέτζιο 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 1 έχω την 2 των γυναικών. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 7, παράγραφο 1, β, μικρό, συμβιβαστική, δι, αγγλική, από τέσσερι πολιτικέ ομάδε. υπέρ, κατά, απόχέ. δεκτή. Άρθρο 8, παράγραφο 5, την 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, απόχέ. απορρίπτεται. 59, Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 59 της κυρίας Παπαδοπούλου. ψηφίζετε; Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 26 υπέρ 17 κατά μία αποχή. Γίνεται δεκτή η 59. Μετά το άρθρο 9 έχω την προφορική τροπολογία Τσέγκορ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Φτάνουμε τώρα σε αιτιολογικές σκέψεις. Θέτω σε ψηφοφορία τις τροπολογίες 18 και 19 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Η 20 έχει αποσυρθεί. Συνεπώς θέτω σε ψηφοφορία την 1 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην αιτιολογική σκέψη 4 έχω την 2, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 εισηγητή, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 24 Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια ψήφος δεκτή. Στην αιτιολογική 8. Έχω την 1 της Ρέτζιο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Μετά έχω την 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχω δύο ταυτόσημες τώρα, την 25 της κυρίας Παπαδοπούλου και την 3 της Ρέτζιο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στην 10, παράγραφος 4 της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην 11, έχω την 3 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στην αιτιολογική 13 την 27 Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά την 13 έχω την 6 της Ρέτζιο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. ψηφίζετε παρακαλώ. 34 υπέρ, 5 κατά. 5 αποχές. Η έκθεση Σόγκορ γίνεται δεκτή. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τον εισηγητή αν θέλει να αφήσει το όνομά του επί της εκθέσεως ή αν θέλει να αφαιρεθεί το όνομά του λόγω του αποτελέσματος. with that, Το έχω συνηθίσει αυτό και στη δική μου χώρα το ίδιο μου συμβαίνει. Alors, euh, je comprends que le rapporteur... Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο εισηγητής θέλει να αφαιρέσει το όνομά του. Όχι, όχι. Ε, επαναλαμβάνει ότι το έχει συνηθίσει ο εισηγητής, αλλά το αφήνει το όνομά του. Λοιπόν, δέχεται και την εντολή διαπραγμάτευση. Συνεπώ, κατά συνέπεια συνεχίζουμε και θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, έκανα λάθος λέει ο Πρόεδρος. Ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Πέραστη ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 13 κατά, 0 οι αποχές. Η νομοθετική πρόταση συνεπώς ε, ε, προωθείται, γίνεται δεκτή. Θα ψηφίσουμε τώρα. Για, ε, για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Euh, Ψηφίσαμε λοιπόν το νομοθετικό ψήφισμα τροποποιημένο. Συνεπώς, η επιλογή η οποία δίδεται τώρα στα μέλη είναι εάν επιθυμούν να ορίσουν την εντολή διαπραγμάτευσης επί τη βάση μιας ψηφοφορίας στην Επιτροπή μας ή θα προτιμούσαν να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να επικυρώσει την συγκεκριμένη εντολή διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Όρη και μετά ο κύριος Θέρκαθ. Η θα προτιμούσα να ζητησουμε απο την ολομελεια να επικυρωσει την συγκεκριμενη εντολη διαπραγματευσης ο κυριος ορη και μετα ο κυριος θερκαθ η συσταση μου θα ήταν, Πρόεδρε, να περάσει στην Ολομέλεια, προκειμένου η Ολομέλεια να επιβεβαιώσει την εντολή την Δευτέρα. Νομίζω ότι είναι σαφής η πλειοψηφία και νομίζω ότι η απόφαση της Επιτροπής μας θα πρέπει να καθοδηγήσει τους διαπραγματευτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, εντολή της Επιτροπής. Κυρία Λάμπερτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί το σύνολο του Κοινοβουλίου και θα προτιμούσαμε να περάσει την Ολομέλεια. Alors nous allons faire un vote sur la procédure. Κοιτάξτε, θα ψηφίσουμε τότε και για τη διαδικασία. Ποιοι επιθυμούν η απόφαση να ληφθεί από την Ολομέλεια. Ποιοι είναι υπέρ της Ολομέλειας, συνεπώς. Ποιοι είναι κατά. Κοιτάξτε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, αυτή η νέα διαδικασία ακόμα είναι σε διαδικασία στρωσίματος. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει απόλυτα. Καταλαβαίνω ότι ο δικός χάρτης έτσι όπως έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων λέγει το εξής θα πρέπει εμείς να ψηφίσουμε για να δούμε αν υπάρχει εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να περάσουμε σε διαπραγμάτευση και η εντολή αυτή θα πρέπει να δοθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελείται από 25 μέλη, τότε αυτόματα θα πάμε στην Ολομέλεια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σας ρωτήσω για το αν θέλετε να κάνετε το ένα ή το άλλο. Η πλειοψηφία η οποία θα προέλθει από την εντολή που θα δοθεί προς την Επιτροπή για την εκκίνηση του τριμερούς διαλόγου θα επηρεάσει άμεσα το τι θα κάνουμε. Εντάξει, να το επαναλάβω. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία η οποία θα μας πει αν θα δώσουμε εντολή στην Επιτροπή να ξεκινήσει επί της συγκεκριμένης βάσεως τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο. Για να είναι έγκυρη η εντολή αυτή απαιτούνται 25 ψήφοι υπέρ. Ο κύριος Σορή έχει ζητήσει μια διευκρίνηση. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει να ψηφίσουμε υπέρ και τι θα ψηφίσουμε κατά. Τι είναι το ναι, τι είναι το όχι. Σας παρακαλώ επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί πρέπει να είναι σαφές. Τι ερωτούμαστε για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, να ξέρουμε τι είναι το ναι, τι είναι το όχι. Αν ψηφίσετε υπέρ με μια πλειοψηφία 25 ψήφων τουλάχιστον, οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν επί τη βάση των αποφάσεων που μόλις ψηφίσαμε. Εάν μία πλειοψηφία των 25 δεν υλοποιηθεί, τότε η εντολή θα πρέπει να δοθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία επί της εντολής διαπραγματεύσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Le vote est ouvert. Il y a un e Il y a un PPE de trop. Quel est le dernier suppléant PPE à être rentré Ποιος είναι ο τελευταίος ε, αναπληρωτής του ΕΛΚ που μπήκε στην αίθουσα. Ησυχία παρακαλώ λέει πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 18 κατά. Συνεπώς η εντολή θα δοθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όχι από την Επιτροπή μας. Ησυχία παρακαλώ. Πριν προχωρήσουμε σας προτείνω να υπάρξει μια διαβούλευση παρακαλώ ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες για να συμφωνήσετε επί τη βάση ποιων τροπολογιών θα κατέβουμε στην Ολομέλεια. Λογικά θα πρέπει οι τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή μας συνολικά να κατατεθούν στην Ολομέλεια και ίσως να υπάρξουν και κάποιες επιπλέον διαπραγματεύσεις. Αλλά αυτά θα τα αποφασίσουν οι πολιτικές ομάδες μεταξύ τους. Φτάνουμε επιτέλους στο σημείο 34. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του συναδέλφου Φιλίπ Μπουλόν για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, να σας πω ότι η τροπολογία 11 έχει αποσυρθεί για να είναι συμβατή με την έκθεση επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Συνεπώς η 11 έχει αποσυρθεί και ψηφίζουμε στην παράγραφο 1, στο άρθρο 1, την 36. Ποιοι είναι υπέρ της 36. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 4 αποσύρθηκε. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 έχω την 37 Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 37. Ψηφίσατε όλοι πέρα στη ψηφοφορία. 16 υπέρ, 24 κατά, δεν γίνεται δεκτή. Άρθρο 4 παράγραφος 3 την 5 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Άρθρο 39 μάλλον είναι συμβατή, ποιοι είναι υπέρ. Για μια στιγμή λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία την 38 της κυρίας Παπαδοπούλου. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 39, συμβατή. Ψηφίζουμε αυτήν τώρα. Υπέρ, κατά αποχής δεκτή. Η 6 αποσύρθηκε. Η 7 επίσης. Έχω την 40 Μαλίκα Μπεναρά Μπατού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο C Έχω την 41 Παπαδοπούλου με μια προφορική τροπολογία. Αντίρρηση δεν υπάρχει. Θέτω σε ψηφοφορία την 41 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο C νέο. Έχω την 8 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Άρθρο 6, παράγραφος 1, έχω την 43 μπουλόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 42 Παπαδοπούλου, συμβατή, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Άρθρο 6, παράγραφος 2, συμβιβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Άρθρο 6, παράγραφος 3, 46, Μαλικά Μπεναραμπατού, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Άρθρο 7 παράγραφος 1 εισαγωγικό τμήμα 47 μπουλόν ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 7 παράγραφος 1 σημείο β μικρό ένθετο 1 48 Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 Μαλίκα Μπενιαραμπατού ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή στο εισαγωγικό τμήμα. Έχω την 50 Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 11 στον τίτλο 2 αποσύρθηκε. Θέτω σε ψηφοφορία την 51 Μπουλόν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Άρθρο 7 επί του τίτλου. Έχω την 52 Μπουλόν και Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 12 αποσύρθηκε. Θέτω σε ψηφοφορία την 53. Μπουλόν Παπαδοπούλου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έχω την 13. Μπουλόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική Β. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή την 10 παράγραφος 1 την 15 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 56 Μπεναράμπα του συμβατή ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 παράγραφος 1 την 16 Μπουλόν υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 συμβατή υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 παράγραφος 2 συμβιβαστική σι αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 παράγραφος 3 συμβιβαστική D αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή άρθρο 12 παράγραφος 4 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή άρθρο 12 παράγραφος 5 τροπολογία 60 Παπαδοπούλου με μια προφορική τροπολογία δεν υπάρχει αντίρρηση θέτω σε ψηφοφορία την 60 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή Άρθρο 12, παραγραφο 5 5α μικρό, 61, Παπαδοπούλου Μπουλόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ δεκτή. Άρθρο 13, 20, Φιλίπ Μπουλόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ δεκτή. Άρθρο 13, 62, Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ δεκτή. Άρθρο 14, παράγραφος 3, συμβιβαστική ή αγγλικό, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Άρθρο 14, παράγραφος 14, 4 αλφα μικρό, 65, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Άρθρο 15, μετά την παράγραφο 1, έχω την 66, Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείωση αγγλικό νέο, 23 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 16, παράγραφος 2, έχω την 67, Μπεναράμπα του. Εδώ έχει ζητηθεί προφορική τροπολογία από τους πρασίνους, δεν υπάρχει αντίρρηση, τίθεται σε ψηφοφορία. Ε, η τροποποιημένη 67, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Άρθρο 16 παράγραφος 3, 68 μπουλό, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 17 παράγραφος 3, 25 μπουλό, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 26 παράγραφος 3, 69 Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 26 Παπαδοπούλου με μια προφορική τροπολογία δεν υπάρχει αντίρρηση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Μετά το 2 έχω την 27 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Μετά το 3 έχω την 28 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στο 5 29 Παπαδοπούλου ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στο 6 1 Μπουλό ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Θέτω σε ψηφοφορία την 30 τώρα, Βλόσοβιτς. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στο 7 την 31 Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στο 9, 32 Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στο 10, οι δύο, Μπουλόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στο 12.33, Παπαδοπούλου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τρία αποσύρθηκε, θέτω σε ψηφοφορία την 34 Βλόσοβιτς. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μετά τη 15 έχω την 35 Τη Ανθής Μακίνταερ. ευχή είναι υπέρ, κατά, υπέρ. Δεκτή. Το σύνολο τώρα της νομοδότησης τίθεται σε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορία. 36 υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές, συγχαρητήρια. Φτάνουμε Πάμε τώρα στην προφορική ερώτηση για τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες. Τροπολογία 1. Αντζελίλη Κώσα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Κίνγκα Γκέντς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα τεσσάρων ομάδων. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, τρο... συμβαστική ΣΕ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το κείμενο ολόκληρο. Ποιο είναι, ε, ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 39 ψήφισαν υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Οπότε η προφορική ερώτηση θα υποβληθεί με αυτή τη διατύπωση στην Ολομέλεια. Και περιμένω από τις ομάδες να γραφούν για συμμετοχή. Σημείο 36 τώρα. γνωμοδότηση του Τόμας Μαν για τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια της Ένωσης και κατάργηση της οδηγίας 96-67 του Συμβουλίου. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε δεύτερη ψηφοφορία για την γνωμοδότηση, μια και η έκθεση επί της ουσίας, στην οποία αναφερόταν η γνωμοδότηση, αναπέμφθη από την Ολομέλεια στην αρμόδια επιτροπή. Οπότε ξανάρχισε η διαδικασία. Ο εισηγητή μα προτείνει να επιβεβαιώσουμε την γνωμοδότησή του που την είχαμε ήδη εγκρίνει το Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, χωρίς αλλαγές. Ας ψηφίσουμε λοιπόν την γνωμοδότηση του κυρίου Τόμας Μαν με τη μορφή που έχει 18 Σεπτεμβρίου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 36 ψήφισαν υπέρ, 7 κατά. Χωρίς αποχές. Οπότε επιβεβαιώνουμε τη γνωμοδότηση που είχαμε εγκρίνει το Σεπτέμβριο ήδη. Και τέλος ψηφοφορίες. Πέραμε λοιπόν στο σημείο 37 το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Τζιν Λάμπερτ με θέμα την πρόσβαση στην περίθαλψη των ευάλωτων ομάδων. Madame la vous avez la parole. Έχετε το λόγο, κυρία Συγγετρία. Και παρακαλώ όσοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα να το κάνουν ε, χωρίς φασαρία. Madame la Uh, Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε. Είσαστε κάποιοι μόνο εδώ σε μια ακρόαση για την έκθεση αυτή πριν από κάποιες εβδομάδες και νομίζω ότι η ακρόαση ήταν πάρα πολύ δυναμική. Η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή. Ε, ακούσαμε διάφορες οργανώσεις που ε, συμμετέχουν στην παροχή ε, υπηρεσιών και φροντίδας σε διάφορες μα μας ε, ενημέρωσαν αρκετά καλά για το τι συμβαίνει στις παρούσες συνθήκε. Η έκθεση που υπέβαλα αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει αρκετά κενά. Πολλά σημεία λείπουν. Εν μέρη, επειδή περιοριζόμαστε σε 6.000 χαρακτήρες και νομίζω ότι εξάλλου βρισκόμαστε στην αρχή μιας ε, τέτοια εργασίας, οι συνάδελφοι ασφαλώς θα έχουν πολλά να προσθέσουν. Η πρόσβαση, μάλλον ε, η, υπογραμμίζουμε θέματα παροχής φροντίδας σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες. Δεν κοιτάμε το συνολικό ζήτημα της ένδυας στην παρούσα φάση ή άλλες πτυχές της ε, φτώχειας υπάρχουν άλλες ε, εκθέσεις για τους άλλους τομείς αυτούς. Μία άλλη έκθεση πραγματεύεται και την κοινωνική στέγαση. Έχουμε και την προφορική ερώτηση σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στην έκθεση αυτή σε θέματα περίθαλψης. Στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς εδώ στην Επιτροπή. Φυσικά η βασική αρμοδιότητα είναι της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και γι' αυτό αναφέρω κάποιες πτυχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής για να μην πούμε στην, στα νερά της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος. τίθονται ε, το θέμα του τι συμβαίνει με τα άτομα που έχουν αναπηρία, με τους πρεσβύτερους, με τα παιδιά που βρίσκονται στα χέρια της δημόσιας ε, φροντίδας. Αυτό αναφέρθηκε και χτες στην πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια από τα θέματα αυτά θα πρέπει να διασαφινιστούν σε ό,τι αφορά τις ε, τάσεις που σημειώνονται, σε ό,τι αφορά το αυξανόμενο κόστος, σε ό,τι αφορά το κόστος ε, των υπηρεσιών για τους πιο ηλικιωμένους. Νομίζω ότι κάτι που απασχολεί την Επιτροπή μα είναι μια μετατόπιση που φαίνεται να υπάρχει σε ό,τι αφορά τα επιδόματα κοινωνική ασφάλιση. Είναι περιοριστική σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στι υπηρεσίε περιθαλψή. Αυτό κατέστη σαφέ και στην ακρόαση και από τι εκθέσει άλλων οργανώσεων. Είναι ότι πολλοί κόσμοι χάνει την πρόσβαση, το δικαίωμα πρόσβαση στην υγειονομική περιθαλψή μετά από κάποια περίοδο που είναι στην ανεργία. Αυτό από προσωπικής άποψης ε, φαίνεται ότι αποτελεί πάρα πολύ σκληρή τιμωρία. Γιατί είναι και μεγάλη ενεργεία σήμερα στην αγορά εργασία, είναι δύσκολο να βρει κανεί δουλειά. Ε, Επίση, ε, κοιτάμε τι νοριακέ καταστάσει, πω ο κόσμο δεν έχει, δεν υπάρχουν εναρμονισμένε υπηρεσίε και υπάρχει ένα κενό σε ό,τι αφορά την παροχή Ε, Ένα άλλο θέμα είναι οι περικοπές που γίνονται. Πολλά κράτη-μέλη φαίνεται ότι έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την παροχή υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, είτε είναι διανετική είτε είναι σωματική αυτή η αναπηρία. Αυτό φαίνεται ότι περικόπτεται, ότι τα πρότυπα, οι προδιαγραφές ε, περιθάλψης ε, πέφτουν. Και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει, δεν θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα άλλα ζητήματα τώρα κάποια άλλα προσκόμματα. Το στίγμα, για παράδειγμα, που συνδέεται με κάποιες ε, ε, παθήσεις, με κάποιες ε, καταστάσεις και διάφορα εγκλήματα που σχετίζονται με το στίγμα αυτό. Δεν θα πρέπει να το σκεφτώ, να το ξεχνάμε αυτό. Και τέλος θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ποιότητα των συνθήκων εργασίας και αυτό επηρεάζει την ε, παροχή ε, υπηρεσιών περίθαλψης. Ε, έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού, με την ποιότητα εκπαίδευση του προσωπικού που παρέχει την περίθαλψη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Τώρα, θα ήθελα να αναφέρω αυτό που είπε και ο Επίτροπος Άντο χτες σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο κόστος της αδράνειας, το μακροπρόθεσμο κόστος του να μην της μη πρόληψης σε ό,τι αφορά και τα άτομα αλλά και τις υπηρεσίες ε, δημοσιονομικής περιθάλψης. Φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές οι οποίες έχουν επιβληθεί εμπεριέχουν και μία απουσία παντελή της μακροπρόθεσμης διάστασης, του τι θα συμβεί, δηλαδή ποιος θα είναι ο αντίκτυπος μακροπρόθεσμα η Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει, για παράδειγμα, ότι η Επιτροπή μας έχει καταστήσει σαφές ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το ΑΕΠ, να δούμε και το κοινωνικό κόστος. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη και να τα λαμβάνουμε υπόψη σε εποχές κρίσης. Επίσης ακούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εγκαταλείπεται η διάσταση της κοινοτομίας και της κοινωνικής ε, κοινοτομίας, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχτεί ότι αυτό αποφέρει κέρδος τα κράτη-μέλη ξαναγυρνάνε στις παλιές συνήθειες και αφήνουν τις νέες ιδέες οι οποίες ε, απέφεραν κέρδος. Επίσης, αύξηση του αποκλεισμού και βλέπω, βλέπουμε ότι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίε περιθάλψη αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Σε ό,τι αφορά τι προτάσει τώρα, συνειδητοποιώ και αντιλαμβάνομαι ότι είναι μετριοπαθεί οι προτάσει μου και είμαι βέβαιη ότι και άλλοι συνάδελφοι θα θέλουν να προσθέσουν προτάσει και προφανώ όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν και στα εθνικά σχέδια μεταρρύθμιση. Τον έφερε άλλωστε και ο Επίτροπο χτε είναι σαφέ εδώ στην Επιτροπή ότι αυτή η κοινωνική πτυχή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις μελέτε αντικτύπου προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα τα οποία λαμβάνουμε από τις χώρες δεν υπονομεύουν αυτές τις πολύ πολύ πολύ βασικές ε, παροχές που τονίζουμε εδώ και χρόνια ότι είναι σημαντικές για για την κοινωνική ε, συμμετοχή, για την αξιοπρέπεια των ατόμων που και προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνική ασφάλεια μεταξύ των κρατών μελών και αυτό έχει να κάνει και με την, με την ε, εφαρμογή τη οδηγία 2048 σε ό,τι αφορά και τους ε, κατοίκου που μένουν σε ένα κράτο μέλο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ε, υγειονομική περιθαλψη, να μην βρεθεί ένα φτηνό υποκατάστατο. Τα χρήματα τα οποία έχουν ως στόχο της ευάλωτη ομάδα θα πρέπει επίση να αξιοποιούνται, γιατί πολλά κονδύλια δεν αξιοποιούνται. Επίσης ανακύπτουν θέματα για το πώς θα διατηρηθούν τα μέτρα υποστήριξης για τους παρόχους του υγειονομικής περίθαλψης και ένα άλλο θέμα που ακούσαμε είναι για το, το ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αναπτύξουν ένα κοινωνικό διάλογο για τις ανάγκες του τομέα. Αυτά αποτελούν λοιπόν τη βάση επί της οποίας ε, θα εργαστούμε. Προφανώς και οι συνάδελφοι θα υποβάλουν και άλλες ιδέες. Προσβλέπω να τις ακούσω και θα ήθελα τελικά να διαμορφωθεί κάτι θετικό, κάτι χρήσιμο στο τέλος της δικασίας αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έπρεπε να, θα, ήθελα να πω ότι δεν έχω πολλά να προσθέσω γιατί η κυρία Λάμπερτεκ μας υπέβαλε μια πολύ καλή έκθεση η οποία ξεκαθαρίζει ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τονίζει πόσο σημαντική είναι τουλάχιστον η πρόσβαση στην περίθαλψη. Και η συγκεκριά επίσης ε, διευκρίνησε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά και το συνεπαγόμενο κόστος. Και φυσικά είναι σημαντικό επειδή μιλάμε για άτομα με αναπηρία, είναι σημαντικό το θέμα της ε, συμπερίληψης, της συμμετοχής, της ε, ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες ομάδες πλήττονται. Τι βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό αυτοί που έχουν δουλειά δεν έχουν κάποιες φορές πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες γιατί πολύ απλά κοστίζουν υπερβολικά. Ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι το πρόβλημα των διασυνοριακών χρηματοδοτήσεων και της ε, διασυνοριακής ε, αποζημίωσης, της αποζημίωσης μάλλον των συνεργειακών υπηρεσιών περιθαλψής. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσει κανείς επιστροφή του κόστους αυτού. Και εδώ σίγουρα θα πρέπει να επέμβουμε. Είμαι πολύ αισιέδειξη ότι μαζί με την Jean Lambert θα καταφέρουμε να καταρτήσουμε μια πολύ σωστή έκθεση. Η κυρία Άρκιν και μετά ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ. Η Τζένι είπε ότι θεωρεί ότι πολλά θα χρειαστεί να προσθετούν σε αυτή την έκθεση. Δεν είμαι σίγουρη. Θεωρώ ότι είναι πολύ συνεκτικό και μεστό το κείμενό τη. Εγώ προσωπικά δεν έχω πολλά να προσθέσω, μια ερωτήσει να κάνω, να προσθέσω μια σκέψεις αν θέλετε. Υποστηρίζω σαφώς ε, την ιδέα ότι δεσμευόμαστε και έχουμε δεσμευτεί στα πλαίσια του ΟΗΕ και των σχετικών συνθήκων για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό περιλαμβάνεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά ε, παρόλα αυτά δεν ανταποκρινόμαστε σε τις δεσμεύσεις αυτές και σε ό,τι αναφέρει για την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, σύμφωνο να ρωτήσω για την σύσταση 17. Αναφέρει τις, τις αντιφάσεις μεταξύ του κανονισμού και της ε, οδηγίας ε, της οδηγίας 2048 ε, και του κανονισμού 883 του 2004. Πώς θεωρείτε ότι μπορούν να λυθούν αυτές οι αντιφάσεις. Επίσης, στην ε, έκθεση αναφέρει ότι κάποια παιδιά δεν εμβολιάζονται, δεν κάνουν τα βασικά εμβόλια. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Έχετε πιο πολλές πληροφορίες να μας δώσετε. Και πάλι συμφωνώ να πω για το ότι θα πρέπει όντως να λαμβάνουν υποστήριξη η πάροχη των υπηρεσιών περίθαλψης. Γιατί αποτελούν ουσιαστικά το μοναδικό δίκτυο ασφαλείας που έχουμε στην παρούσα φάση. Ιδιαίτερα σε όταν αφορά και τις οικογένειες των ε, ατόμων με προβλήματα. Στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να ε, χρησιμοποιούν ε, επιμέρους στόχους για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες αυτές ομάδες. Και αυτοί οι επιμέρους στόχοι θα μας επέτρεπαν να καταλάβουμε την πλήρη έκταση της κρίσης και του αντίκτυπου της κρίσης στους πλέον ευάλωτους. Πολλές φορές το έχουμε πει εδώ στην Επιτροπή μας ότι χρειαζόμαστε κοινωνική επιτήρηση ε, σε ό,τι αφορά τις χώρες που συμμετέχουν σε προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπέκερ. Και μετά, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, ωραία. Ο κύριος Μπέκερ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Όντω είναι πάρα πολύ επαγγελματική η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Κάποιες πτυχές να υπογραμμίσω και ίσω να κάνω και κάποιες τροπολογίες. Αλλά πρόκειται για θέματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Καταρχάς, όντω θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πλέον ευάλωτες ομάδες, όχι στο σύνολο, στο συνολικό φάσμα των θεμάτων που εμπλέκονται. Όχι, να εστιαστούμε στις ευάλωτες ομάδες. Να υπογραμμίσω επίσης πόσο σημαντική είναι αυτή η ανεπίσημη φροντίδα, ιδιαίτερα από την οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το αντιληφθούμε, να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που α, αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά. Επίσης, να κοιτάξουμε τη μακροπρόθεσμη ε, περίθαλψη. Και σε αυτή να λεφτή υπόψη ε, η πάροχη αυτή της φροντίδας. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η έκθεση. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα ήθελα να λάβει το λόγο. Όχι, ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πολύ τους συναδέλφους. Πολύ θετικά τα σχόλια τους. Και ακόμα και από τα σχόλιά σας πρέπει να πω ότι παίρνω ιδέες πολύ χρήσιμες. Κάποια ερωτήματα μου τέθηκαν. Καταρχάς για τα βασικά εμβόλια. Από πού ήρθε τα στοιχεία γιατροί του κόσμου, από μια έκθεση των γιατρών του κόσμου. Για την Ελλάδα τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, ξέρω ότι το έχουν θίξει και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, αλλά και για τα εμβόλια του εμβολιασμού στην Πορτογαλία. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και στο δικό μου κράτος μέλος ε, κάποιες ομάδες ε, δεν ε, πιάνονται, αν θέλετε, στο κοινωνικό δίκτυο. και σίγουρα σε χώρες όπου ο κόσμος πρέπει να πληρώσει για το κόστος αυτών των βασικών εμβολίων. Είναι πραγματικά τρομακτικό, έχετε δίκιο. δεν λαμβάνει και υπόψη αυτή η πολιτική του στόχους που έχουμε θέσει για τους εμβολιασμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, ε, διαφορές και τις αντιφάσεις μεταξύ του κανονισμού και της ε, οδηγίας ε, για την διασυνοριακή υπερίθαλψη και για τους μακροπρόθεσμους κατοικούς. Το θέμα λοιπόν είναι από ποιο σημείο μπορεί κανείς να έχει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη. Εκεί υπάρχει αντίφαση μεταξύ κανονισμού και οδηγίας. Αυτό ανακύπτει ως ε, ολοένα και πιο μεγάλο θέμα σε διάφορα Αν και δεν το αναφέρουν αυτό ίσως ε, επισήμως. Και το ακούμε και στις συνεδριάσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολίτη. Επίσης, ε, ενδιαφέρουσα ιδέα για την κοινωνική επιτήρηση. Να δω και τις ε, τροπολογίες σας. Νομίζω ότι θα είναι πολύ επικοδομητική τελικά η εκθέση. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, λοιπόν. Ωραία. Θαυμάσια. «28 Φεβρουαρίου το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Θα τις εξετάσουμε στις 20-21 Μαρτίου ε, τις συμβαστικές τροπολογίες της 29 Μαΐου και θα ψηφίσουμε την επαύριο 30 Μαΐου για να διαβιβάσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια της Δευτέρας Ιουλίου. Ε, στην έκθεση του, στην Ολομέλεια του Ιουλίου, συγγνώμη. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και προχωράμε στο επόμενο, το 19, που κανονικά προβλεπόταν για χθες, αλλά έγινε μια αντιστροφή των σημείων. Οπότε θα εξετάσουμε τώρα το σημείο 19 και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και την εξέταση των τροπολογιών της έκθεσης της κυρίας Γιαζοβίετσκα με θέμα την επιβολή της οδηγίας 7196 για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Ε, ε, ε, de Euh, Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Γιαζοβιέτσκα, για να μας ε, υποβάλει τα πρώτα της σχόλια για τις 833 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την έκθεσή της. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ζητώ, που, ζητώ συγγνώμη που χθε ζήτησα την αντιστροφή αυτών των σημείων και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Γραμματεία και τους συναδέλφους που το δέχτηκαν. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους ε, ε, που κατέθεσαν τροπολογίες. Όπως είπε και η, Πρόεδρος, ε, κατατέθηκαν πάνω από 800 τροπολογίες, κάτι που δείχνει την, το τεράστιο ενδιαφέρον που προκάλεσε η έκθεση αυτή. Φυσικά θα καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες, αλλά και για τη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να προστατεύσουμε τους αποσπασμένους ε, ε, εργαζομένους και φυσικά να τηρήσουμε τους στόχους της οδηγίας 96-71 για το θέμα αυτό. Ε, υποχρέωσή μου στην αναζήτηση συμβαστικών τροπολογιών είναι να προτείνω λύσεις ε, που θα είναι πολύ σημαντικές ε, για την προστασία των εργαζομένων, όπως είπαμε και με τους κοιόδης ηγητές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδηγία θα πρέπει να βοηθήσει την εφαρμογή την, ε, και την εκτέλεση των υποχρεώσεων της βασικής οδηγίας ε, του 96 που μιλά για την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Για να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε στην εφαρμοστική οδηγία σαφείς ε, διαφανεί διατάξει ε, και που δεν θα είναι αντιφατικέ με τι ήδη δεσμευτικέ διατάξεις που ισχύουν από τη βασική οδηγία. Όλε οι πολιτικέ ε, ομάδε δηλώνουν, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι ο υπέρτερο στόχο τη οδηγία αυτή είναι η εξασφάλιση και η διεύρυνση τη προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. Είμαι πεπισμένο ότι η οριστική έκθεση, το οριστικό κείμενο θα είναι ισορροπημένο και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σημείο αφετηρίας για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να στηριχτούμε σε μια ορθολογική θέση, μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις και λύσεις με τον συνομοθέτη. Η ΔΕΜΗ ελοχεύει ο κίνδυνος να μπλοκαριστεί αυτό το σχέδιο, κάτι που θα είναι η χειρότερη δυνατή εξέλιξη για τους αποσπασμένους εργαζομένους, γιατί έτσι δεν θα έχουμε εισαγωγή των διατάξεων που θα βελτιώνουν την κατάστασή τους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Πριν μιλήσω για τις τροπολογίες, θα ήθελα να επισημάνω κάποια βασικά σημεία που θα τα λάβω υπόψη και στην επεξεργασία των ε, συμβαστικών τροπολογιών. Καταρχήν θέλουμε ε, λογικά και ισορροπημένα μέσα ε, για την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. Θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες ό,τι αφορά τους όρους πρόσληψης και μάλιστα οι πληροφορίες είναι προσιτές και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Τρίτον, θα πρέπει να εναρμονιστεί το θέμα της απόσπασης και τα διάφορα στοιχεία. Επίσης, ε, πρόσβαση στην πληροφορία των ρυθμιστικών αρχών. Πέμπτον, θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. Για όλα αυτά τα σημεία μιλήσαμε στις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και θα ε, τα υποστηρίξω ιδιαίτερως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες τροπολογίες, θα ήθελα να ξεκινήσω από, τις, ε, από την πρόταση με την οποία μιλούμε για την ίση ε, ε μεταχείριση των αποσπασμένων με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Συμφωνώ με την ε, πρόταση του άρθρου 3 της οδηγίας 9671 στην οποία αναφέρεται η ε, αναφέρονται οι διατάξεις της οδηγίας της χώρας υποδοχής, ε, οι οποίες θα ισχύουν και για, τις, ε, για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, στην περίπτωση μόνο που είναι όμως ευνοϊκότερες από τις διατάξεις της χώρας προέλευσης. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 221, 222, 227, μιλούμε για τα θέματα των αποσπασμένων εργαζομένων και την παροχή των υπηρεσιών αλλά με τις προτάσεις αυτές θα, θα οδηγηθούμε στην ε, ε, διαγραφή τέτοιων ε, διατάξεων προστασίας που κανονικά θα έπρεπε να ισχύουν. Πολύ συχνά η απόσπαση των εργαζομένων λαμβάνει χώρα σε οικονομικούς τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη εργαζομένων στη χώρα υποδοχής. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο ερωτηματικό για τη θέση εργασίας περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων φαίνεται ότι η απόσπαση εργαζομένων γίνεται κυρίω από τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι περίπου 70% των αποσπασμένων εργαζομένων προέρχεται από χώρε παρόλα αυτά τη Δυτικής Ευρώπη. και κάθε χρόνο 220.000 έχουμε από την ε, Γαλλία και 180.000 ε, από τη Γερμανία. Όπως είπα επανειλημμένως, θεωρώ ότι η βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες για τους εργοδότες και εργαζόμενους είναι ε, κομβικό σημείο της εφαρμοστικής οδηγίας. Και χαίρομαι που το θέμα αυτό έτυχε ευρείας υποστήριξης και από τους ευρωβουλευτές αλλά και από τους κοινωνικούς μας εταίρους. Ένα απαραίτητο άλλο σημείο είναι ότι σε κάθε χώρα μέλη θα υπάρχει ένα και σίγουρο μέσο και μια σίγουρη πηγή ε, πληροφόρησης. Single National Official Website, μία ενιαία ιστοσελίδα, ένας ενιαίος ιστότοπος, γιατί μόνο όταν έχουμε μία πηγή πληροφοριών θα δημιουργηθεί μία διαφάνεια και μία σαφήνεια. Και έτσι διευκολύνονται και όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Ακόμη και η διεύρυνση αυτών των πληροφοριών θα πρέπει ε, να προέρχεται από ένα και μόνο μέσο, από μία πηγή. Και μάλιστα αυτή η πηγή θα είναι εθνική. Όταν λέμε national δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την ειδική κατάσταση των ομοσπονδιακών ε, κρατηδίων ή κάποιων αυτόνομων περιφερειών. Πρέπει να είναι επίσης επίσημη αυτή η ιστοσελίδα. Αυτό λέμε official. Θα... Έτσι θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνει. Το... Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το θέμα των γλωσσών. Ε, σε διάφορες γλώσσες, σε ποια γλώσσα θα πρέπει να, να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε σε ποιες γλώσσες θα πρέπει να μεταφράζονται αυτές οι πληροφορίες. Ε, σχετικές τροπολογίες κατέθεσαν η κυρία Χίρς, ο κύριος Μπρόκ, ε, η τροπολογίες 432, 33 κτλ. Πιστεύω ότι θα πρέπει για το θέμα της γλώσσας να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή ε, λύση για τους εργοδότες και για τους ε, εργαζόμενους. Προτάθηκε και η δημιουργία κέντρων πληροφοριών για τους εργαζόμενους. Η Γιούτα Στάινμπρουκ και ο Στίβεν Χιούς κατέθεσαν τέτοια τροπολογία, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, η Μάρτιν Κάσλερ για παράδειγμα 457, 458, 460 τροπολογίες αναφέρονται στα σημεία αυτά. Όπως και η τροπολογία μου 522. Είχα συναντήσεις με ανθρώπους που εργάζονται σε τέτοια γραφεία επαφή και θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμη η δραστηριότητά τους. Επίσης θεωρώ ότι με την εφαρμοστική αυτή οδηγία δεν θα πρέπει να προβλέψουμε την ε, υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν τέτοια σημεία επαφής. Γιατί σε ορισμένες ε, χώρες έχουμε ελάχιστε τέτοιε περιπτώσει ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις απόσπαση εργαζομένων ή σε πολύ συγκεκριμένου τομεί. Οπότε δεν έχει νόημα σε αυτέ τι χώρε με τόσο περιθωριακό το φαινόμενο τη απόφαση να προβλέψουμε την υποχρέωση δημιουργία τέτοιων γραφείων. Είναι υπερβολική και περί υποχρέωση. Είναι σημαντικό οι ίδιοι εργοδότες να είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους ε, που θα αποσπαστούν σε αυτούς για ε, τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της απόσπασης. Επίσης, ε, θα πρέπει ο εργολάβος να ενημερώνει τον υπεργολάβο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Και η τροπολογία 456 που προτείνει κάτι τέτοιο, ελπίζω να εγκριθεί από την Επιτροπή μας. Στο άρθρο 3 της οδηγίας για την εφαρμογή αναφέρονται δύο κατάλογοι στοιχείων που καταλήγουν στην αξιολόγηση του κατά πόσο ο εργοδότης πληρεί τις διατάξεις ή αν όντως είναι προσωρινή απόσπαση. Αναφερόμαστε καταρχήν στο χαρακτήρα των καταλόγων και την, τον προαιρετικό ή τον δεσμευτικό τους χαρακτήρα. Επίσης, στο κατά πόσο θα πρέπει η κατάλογη αυτή να είναι κλειστή ή ανοιχτή, αδεικτική ή εξαντλητική. Επίσης, η, ανοιχτη αδεικτικη η εξαντλητικη επισης οι τροπολογίες περιλαμβάνουν κάποιε αλλαγέ των στοιχείων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο θα εκτιμούνται αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των καταλόγων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί η διατύπωση μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου με βάση την η νόμιμη απόσπαση της οδηγίας, της, με βάση την αρχική οδηγία θα απαγορεύεται με βάση την εφαρμοστική οδηγία εξαιτίας της μη τήρησης ενός μόνο στοιχείου του καταλόγου. Προσοχή λοιπόν. Φυσικά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις εκ μέρους των εργοδοτών, αλλά να μην ε, οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου εξαιτία μια ακατάλληλη ε, διατύπωση ή περιοριστική εφαρμογή ε, των κριτηρίων εμποδίζουμε τους εργοδότες να προβούν σε νόμιμες αποσπάσεις εργαζομένων. Επίσης, προσοχή στα κριτήρια. Έχουμε τις τροπολίες 390, 302, 403. Εκεί αναφερόμαστε στον προαιρετικό χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη θα πρότεινα το χώρος, η χώρα προέλευσης και η χώρα υποδοχής να συνεργαστούν προκειμένου να προσδιορίσουν τα στοιχεία που με βάση τον κανονισμό θα ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 90. Ε, το 1996 το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο κατέληξαν ε, στην διαμόρφωση των δικαιωμάτων για τους αποσπασμένους και αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε σήμερα και χαίρομαι ε, που θέλουμε ένα σωστό και διαφανές δίκαιο προκειμένου να μην τροποποιήσουμε τις διατάξεις της αρχικής οδηγίας. Στην οδηγία του στην οδηγία του 96 δεν προκύπτει υποχρέωση ε, εξασφάλισης και μεταφοράς ε, ε, διανυκτέρευσης ή στέγασης και διατροφής των αποσπασμένων εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση καταβολής αυτών των δαπανών, ή την εξασφάλιση επιστροφής αυτού του κόστου, αυτού του κόστους ε, διαμονής, διατροφής και αποζημίωσης, αυτό το καθορίζει το κράτος ε, υποδοχής. Τώρα, αν θα πρέπει να έχω μία ελάχιστη, ε, ελάχιστη αποζημίωση, αυτό ε, καθορίζει το κράτος υποδοχής. Αυτό το προβλέπει η Οδηγία 100. Σε ό,τι αφορά την Οδηγία του 96, που αποτελεί την βασική νομοθετική πράξη, έγιναν δεκτές κάποιες οδηγίες για το, τη διάρκεια εφαρμογής των δικαιωμάτων. Οι οδηγίες, ε, η τροπολογία 397 ε, αντιβαίνει στην αρχή αυτή. Επίσης, ό,τι αφορά το κατάλογο των στοιχείων ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν από τον ε, προσλαμβάνονται εργοδότη. Τέτοιου είδου μέσα και κατάλογοι τέτοιου είδου μέσων θα πρέπει να είναι κλειστή, εξαντλητικοί. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να εξασφαλίσουμε ε, το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα μέσα ελέγχου του άρθρου 9 και να τα διαφοροποιήσουμε από την επιθεώρηση του άρθρου 10. Δηλαδή, να μην περιορίσουμε τον αριθμό των υποθε... επιθεωρήσεων, αλλά απλώ ε, να προσδιορίσουμε τι μπορεί να απαιτεί ο επιχειρηματίας στη διάρκεια της επιθεώρησης, στη διάρκεια της απόσπασης. Πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό το διαχωρισμό. Γιατί ε, επειδή αν πούμε ότι είναι κλειστός ο χαρακτήρας του άρθρου 9, δεν σημαίνει ότι περιορίζουμε τους ελέγχους, αλλά στις πληροφορίες για τα πιθανά μέσα αλλά δίνονται πληροφορίες για τα μέσα ελέγχου. Θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να είναι διαφανής. Έτσι εξασφαλίζουμε και την προστασία και την ασφάλεια των αποσπασμένων εργαζομένων. Το επιχείρημα για τον κλειστό κατάλογο ε, δίνει την δεν δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους να παρακάμψουν αυτή την οδηγία όπως λένε μερικοί. Όπως φαίνεται από εμπειρίες που έχουμε, ένας ε, που ε, εργοδότης που ούτως ή άλλως είναι ανέντιμος δεν θα τηρήσει ούτε τις βασικές διατάξεις της οδηγίας. Αντίστοιχα, ο έντιμος εργοδότης ζητά και δίνει τις πληροφορίες που απαιτεί η οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία να σεβαστεί τα δικαιώματα των αποσπασμένων. Σε όλες τις συζητήσεις και στα έγγραφα λέμε ότι για ενισχύσουμε την οικονομία θα πρέπει να περιορίσουμε το, τη γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθος για τους εργοδότες. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να πριτανεύσει η κοινή λογική. Γιατί η εφαρμοστική οδηγία, μην ξεχνούμε, αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, μία, ένας ανοιχτός κατάλογος και υποχρεωτικός στο άρθρο 9 θα δημιουργήσει τεράστια βάρη και υποχρεώσεις. Η εφαρμοστική οδηγία απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη και σε εκείνα όπου ε, έχουν ελάχιστες περιπτώσεις ε, απόσπασης εργαζομένων. Οπότε από αυτή την άποψη θα πρέπει να υιοθετηθούν διατάξεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στα κράτη-μέλη και τις διαφορές μεταξύ τους. Ούτε θα πρέπει οι διατάξεις οδηγίες αυτές να αντιβαίνουν σε μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η αρχή της αναλογικότητας. Γι' αυτό και δεν μπορώ να δεχτώ τις οδηγίες 5.22 με 5.54 γιατί με βάση τις οδηγίες αυτές ε, η εισαγωγή όλων των μέσων ελέγχου της οδηγίας ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Διαφωνώ με την πρόταση αυτή για υποχρεωτική εφαρμογή όλων των μέσων ελέγχου σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πιο επίμαχο άρθρο της οδηγίας, ε, το άρθρο 12, που μιλάει για την ε, αλληλέγγυη ευθύνη, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είμαι κατά αυτής της πρότασης. Αντίθετα, ε, πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος εκεί που εξασφαλίζεται σωστή προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δυστυχώς ακόμη και στις 8 από τις 27 χώρες που υπάρχει αλληλέγγυη ευθύνη, μόνο στα μισά κράτη μπορεί να εκτελείται απέναντι στον εργοδότη υποχρέωση αυτή. Μετά από ανάλυση λοιπόν της κατάστασης θεωρώ ότι η προσθήκη της διάταξης αυτής όπως προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το στόχο μας που είναι να δώσουμε στους αποσπασμένους εργαζόμενους περισσότερα δικαιώματα. Και μάλιστα ο θεσμό τη αλληλέγγυα ευθύνη με τη μορφή που τον προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα βοηθήσει του αποσπασμένου σε κάθε περίπτωση και όταν έχουν εξαπατηθεί από του εργοδότε να ασκήσουν τα δικαιώματά του. Αν λοιπόν το άρθρο 12 έχει ως στόχο την προστασία των εργαζομένων, θα πρέπει πραγματικά ε, να ε, προστατεύσει τους αποσπασμένους εργαζομένους και όχι αυτούς που εικονικά έχουν προσληφθεί. Γιατί με την κατηγορία αυτή δημιουργείται πρόβλημα. Επίσης, ε, η θέσπιση της αλληλέγγυας ευθύνης μόνο για τις, ε, επιχείρησεις, ε, για τις επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένων θα έχει δυσανάλογα χαρακτήρα και επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Γιατί θα γίνεται ε, θα δίνεται η δυνατότητα ε, γης ε, των πιο δυσμενών διατάξεων, δηλαδή εκείνων στις οποίες ισχύει η αλληλέγγυη ευθύνη. Οπότε η πρόταση τη αλληλέγγυης ευθύνη με τη μορφή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπερβολικά προστατευτικό χαρακτήρα. Οπότε αν εγκριθεί θα διαταράξει την αρχή της ενιαίας αγοράς και μάλιστα θα περιορίσει de facto το, την απόσπαση των εργαζομένων. Γι' αυτό θεωρώ ότι η εφαρμοστική οδηγία θα πρέπει αφενός να περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις ε, που θα προστατεύουν ε, εμπράκτους τα δικαιώματα των εργαζομένων των αποσπασμένων, αλλά θα πρέπει να αφήνει στα κράτη-μέλη τη διακρατική ευχέρεια, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Τέτοιοι μηχανισμοί ε, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους εργοδότες σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Από αυτή την ε, άποψη συμφωνώ με τις 711 ε, ε, Χίρς και 704 Φιλμπένιον. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροπολογίες στη διατύπωση του άρθρου 11, όπως λέω στις τρεις μου τροπολογίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθεί και η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση, την αποτελεσματική εξακρίβωση των καταχρήσεων και την ε, κύρωση σε περίπτωση τέτοιων καταχρηστικών συμπεριφορών. Οι συγκεκριμένες τροπολογίες ε, θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής αλλά θα πρέπει να υπάρχει και αρμονική συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών. Μόνο έτσι θα διευρύνουμε αποτελεσματικά την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων και θα εξασφαλίζουμε ε, στους έντιμους εργαζόμενους τη δυνατότητα ε, ε, αξιοποίησης των δικαιωμάτων που ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι σχετικές τροπολογίες του Τόμας Μαν δείχνουν την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διοικητική συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που κατέθεσαν τόσες πολλές τροπολογίες και να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις ηγητές γιατί συνέβαλαν στο να βρούμε τις καλύτερες νομικές διατάξεις. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε ψήφισε η Επιτροπή ΙΜΚΟ τη γνωμοδότηση για την εφαρμοστική οδηγία και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή αυτή για την πολύ αξιόλογη γνωμοδότηση. Προκύπτει από τις πληροφορίες που έλαβα ότι η γνωμοδότηση και η οριστική της μορφή αποτελεί καρπό μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης και συνεργασίας. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση αυτή θα αποτελέσει καλή αφετηρία και για τη συζήτηση στη δική μας Επιτροπή. Λυπούμε που η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ανέβαλε για το Μάρτιο την ψηφοφορία της δικής της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ και περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για αυτήν την μεγάλη παρουσίαση που έκανα. Τα 20 λεπτά στα οποία μιλήσατε ήταν χρήσιμα πάντως αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω παρακαλώ να μην μιλήσετε για τόση πολλή ώρα γιατί θα ακουστούν μόνο δύο από τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνω ότι έχει ήδη ευχαριστήσει η συγγήτρια του σκιώδης εισηγητές, αλλά φοβάμαι ότι η συνεργασία τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, να σας πω ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο.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 Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εισαγωγή που μας έκανε. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι της πήρε 20 λεπτά να κάνει την εισαγωγή, γιατί είναι πάνω από 800 οι τροπολογίες και πολύ μεγάλη η γκάμα των θεμάτων που κάλυψε. Χαίρομαι για τη δουλειά που έκανε και ξέρω ότι προσπαθεί να προετοιμάσει για το άρθρο 4 ε, για το άρθρο 5 συμβάσεις για το άρθρο 4 λοιπόν, το άρθρο 5 για την ε, βελτίωση της πρόσβασης της πληροφορίας και ήταν πάρα πολύ σαφής εξ αρχής. Για το άρθρο 6 για την αμοιβαία αρρωγή, για το 7 για την ρόλο των κρατών μελών, για το άρθρο 8 για τα συνοδευτικά μέτρα και το άρθρο 9 για τα συστήματα πληροφόρησης. Ε, για όλα αυτά τα σημεία έχει υποβάλει κείμενα. Είναι λοιπόν μια αρχή για μια πολύ σημαντική διαδικασία. Είναι σημαντικά λοιπόν τα θέματα αυτά, αλλά δεν είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Το είπε και η ίδια η συγγήτρια τα άρθρα τα οποία είναι κρίσιμα πραγματικά. Το άρθρο 1 για το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, το άρθρο 3 το οποίο εκτεταμένα το ανέφερε για την πρόληψη καταχρήσεων και της ε, παράκαμψης της οδηγίας, πολύ σημαντικό θέμα, το άρθρο 9 για τα μέτρα εθνικού ελέγχου και τα αμφιλεγόμενα ζητήματα κατά πόσον χρειαζόμαστε ανοιχτή ή κλειστή λίστα. Είναι διαφορετικέ οι απόψεις που επικρατούν ακόμα και στο εσωτερικό των ομάδων και το άρθρο 12 όπως είπε και η συγγήτρια, για το βασικό ζήτημα της ε, της ολόκληρων ευθύνη, την υπεργολαβία. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα, δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία στο ιστορικό των ομάδων. Έχετε δίκιο, είναι δύσκολα θέματα αυτά, περίπλοκα θέματα και θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι παρά το γεγονός ότι έχετε συγκεκριμένες ιδέες, έχουν καταθέσει τροπολογίες και μέλη της ομάδας σας, αλλά και μέλη άλλων ομάδων. Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετό υλικό για να ξεκινήσει μια διαδικασία έβρεσης συμβιβασμού για τα κρίσιμα αυτά θέματα. Είχαμε μια ανταλλαγή ε, αλληλογραφίας την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να παραστώ στην ε, συνεδρίαση των σκιωδών. Δεν θεωρούσα όμως ότι η συνεδρίαση αυτή θα κάλυπτε τα βασικά ε, ζητήματα. Θα προτιμούσα να ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά ζητήματα, άρθρο 1, 3, 9, 12, για να δούμε τι πρώτα μπορούμε να σημειώσουμε σε αυτόν τον τομέα. Να λύσουμε πρώτα τα δύσκολα και μετά νομίζω πολλά θα πάρουν τον δρόμο τους. Ίσως να μην τα καταφέρουμε και ίσως τελικά να, είμαστε, να καταλήξουμε σε διαφορετικές ε, τοποθετήσει. Αλλά θεωρώ ότι καταρχάς θα πρέπει να ψάξουμε συμβιβασμού σε αυτά τα δύσκολα ζητήματα και θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά γρήγορα αν θέλουμε ένα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Επιτροπή και να χρησιμοποιήσουμε και την, ε, τις ευνοϊκές ε, Συνθήκε τη Ιρλανδική ε, Προεδρία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες και να μιλήσω για άλλα 20 λεπτά κι εγώ. Δεν βλέπω τι νόημα έχει. Νομίζω ότι καλύτερα να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι προτιμώ να λύσουμε τα δύσκολα τα ζητήματα και όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τον δρόμο του θεωρώ. Ευχαριστώ. και μετά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητριά. Είχαμε και κάποιες προκαταρτικές συναντήσεις και καταλαβαίνω τι προσπάθεια έχει ήδη καταβάλει και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ διχασμένες οι απόψεις. Πέντε σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Έχω καταθέσει και σχετικέ τροπολογίε. Καταρχά, ε, στο θέμα του ελέγχου. Ένα θέμα του είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Γερμανία, προκειμένου η έλεγχοι να είναι τουλάχιστον ε, τόσο εκτενείς όσο είναι σήμερα, να παραμείνουν τόσο εκτενείς όσο είναι σήμερα. Δεύτερο θέμα, οι εθνικές ιστοσελίδες ως πηγή πληροφορίας, πληροφοριών. Το συζητήσαμε και αυτή την εβδομάδα. Για μας τους φιλελευθέρους έχει νόημα να υπάρχει μια τέτοια ιστοσελίδα όπου ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, αυτός που ψάχνει εργασία, μπορεί να πάρει πληροφορίες, θα ξέρει ότι είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται. Θα βρούμε κάποια κατάλληλη διατύπωση σε ό,τι αφορά το homepage αυτό. Πρόκειται για ένα, θα πρέπει να είναι ένα κεντρικό μέσο το οποίο να εμπιστεύεται ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα για όσους ψάχνουν τέτοιες πληροφορίες. Και θα πρέπει να διατίθενται αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, οι γυριστέ λίστες. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα στο πλαίσιο των φιλελευθέρων. Αν υπάρξει ανοιχτή λίστα, όντως θεωρώ ότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, τα κράτη-μέλη να βάλουν τελικά ό,τι θέλουν στη λίστα και τελικά να εξαιρέσουν κάποια ε, δίκτυα. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό κάπως κλείνουμε μάλλον προς μια κλειστή λίστα. Να υπάρχει μια συγκρισιμότητα, μια ασφάλεια. Αν θέλει μια επιχείρηση, επιχείρηση να δραστηριοποιείται ε, σε διάφορες χώρες. Να ξέρετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές λίστες. Ωστόσο, έχουμε λάβει και τροπολογίες για να συμπεριληφθούν επιπλέον έγγραφα στις κλειστές λίστες. Για το άρθρο 12 τώρα. Και εμείς κάναμε μια σχετική συζήτηση. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι πολύ διχασμένες οι απόψεις και στη Γερμανία. Έχουμε μια από κοινού ευθύνη και είναι καλέ οι που έχουμε. Ξέρω ότι αυτό δεν υπάρχει ωστόσο σε κάποια άλλα κρατημέλη. Γι' αυτό καταθέσαμε την τροπολογία 711 και κάνουμε μια συμβαστική πρόταση, η οποία έχει να κάνει το εξή. Να διατυπώσουμε τους στόχους σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές εισφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρώνονται, αλλά να επαφείται στο κράτος μέλος το πώς θα το διασφαλίσει αυτό, είτε με από κοινού ευθύνη, είτε χωρί αυτήν. Αυτό να επαφείται στα κρατημέλη. Απλά να, ορίσουμε, τον στόχο. Τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω, το θέμα των γλωσσών. Και εδώ υποβάλαμε τροπολογίες που έχουν ε, να κάνουν με τις γλώσσες. Την 431 συγκεκριμένα καταθέσαμε. Κοιτάμε. Το βασικό πρόβλημα, το βασικότερο πρόβλημα μάλλον για έναν εργαζόμενο είναι να μην καταλαβαίνει τις πληροφορίες που έχει. Θα πρέπει λοιπόν να έχει τις πληροφορίες αυτές στη γλώσσα της χώρας από την οποία έρχεται, αλλά και στη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να ε, εργαστεί και στα αγγλικά βέβαια, γιατί είναι η γλώσσα εργασίας πολύ απλά. Είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα της γλώσσας, γιατί αν δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι τα δικαιώματά μου, τι νόημα έχει να τα έχω. Αυτά από πλευράς ε, των φιλελευθέρων. Πολύ βασικό θέμα αυτό για μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ενημερώσω για την ψηφοφορία στην ε, ΙΝΚΟ. Λέει η κυρία Τούρνεν θέλω να σας ενημερώσω για αυτή την ψηφοφορία. Και η κυρία Σρότερ θα μεταφέρει τις απόψεις της ομάδας μετά. Πάντως θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενιαία αγορά, όπως επίσης και για την εμπιστεσύνη που θα πρέπει να δείχνουν οι πολίτες προς την ενιαία αγορά ότι θα σέβεται τα δικαιώματά τους. Η ψηφοφορία ήταν αμφίροπη γενικά. Εγώ σαν εισηγήτρια δεν μπορούσα τελικά να υποστηρίξω τη δική μου έκθεση και ντρέπομαι γι' αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταλήξαμε σε συμβιβαστικές λύσεις εκτός από το 9 και το 12. Πρέπει να τα προσέξετε αυτά γιατί θα καταλήξετε στην ίδια κατάσταση. Πάντως ε, καταλήξαμε σε ενδιαφέρουσες συμβιβαστικές λύσεις ε, για το πεδίο αναφοράς και για την ενιαία αντιμετώπιση, δίκαιη αντιμετώπιση και μεταχείριση στο άρθρο 1, στο άρθρο 3. Υπήρξε μια καλή συμβιβαστική λύση για ένα ανοιχτό κατάλογο των ορισμών. Έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση. Στο άρθρο 5 Εντάξει, στο 6 υπήρξε μια νέα εφεύρεση για την αμοιβαία βοήθεια και ε, σύνδρομη και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος name and shame όπου θα ονοματίζουμε και θα κατηγορούμε τα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται. Αυτό αν θέλετε είναι ένα νέο σημείο στο οποίο καταλήξαμε. Τώρα στο 18 καταλήξαμε σε μια καλή συμβιβαστική λύση σαν το IMI, σαν βασικό μέσο επικοινωνίας, αλλά καταλήξαμε και στη συνέχεια των συμφωνιών που είναι αυτή τη στιγμή σε ισχύ. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Για το 9 σαν παράδειγμα, εμείς ζητήσαμε ένα κλειστό κατάλογο, αυτό ήταν κρίσιμο αλλά και κόκκινη γραμμή για μένα και να το σχολιάσω γιατί σε αυτό αναφέρθηκε και η Νάντια. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Το να δημιουργήσει κανείς νομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κλειστό κατάλογο είναι παρανοϊκό. Δεν επιτρέπει καμία δυνατότητα ευελιξίας. Εγώ αυτό το οποίο πρότεινα σαν εισηγήτρια είναι να πούμε δύο πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει ανοιχτός κατάλογος υπάρχει δυνατότητα αλλαγών και υπάρχει επίσης δυνατότητα να είναι διαφανής η διαδικασία. Αυτό είναι κρίσιμο έτσι ώστε οι πολίτες ας πούμε όταν πηγαίνουμε στη Γερμανία να ξέρουν τι τους περιμένουν, να ξέρουν τι ακριβώς μέτρα ελέγχου θα υπάρχουν και όχι να περιμένουν κάθε φορά για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία μπορεί να χρειάζεται αιώνες για να αλλάξει. Λοιπόν, ε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν κατ' εμέ παρανοϊκό. Δεν ε, μπορώ να στηρίξω την έκθεσή μου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο πλευρές για τον τομέα της οικοδομής είναι υπέρ ενός ανοιχτού καταλόγια. Ακόμα και το Business Europe Χθε πριν από την ψηφοφορία μας έστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι είναι μια καλή λύση αυτή την οποία είχα προτείνει συμβιβαστική. Εγώ είχα πει ότι θα πρέπει να είναι η λύση αναλογική και οι διαθεσιμότητες ε, θα ήταν επίσης ε, δυνατές. Αλλά δυστυχώς υπήρξε ε, θα έλεγα ένα μπλοκάρισμα ιδεολογικού τύπου το οποίο οδήγησε σε αυτό που οδήγησε. Τώρα στην κοινή ανάληψη ευθύνη. Αυτό δυστυχώς δεν πέρασε στην Ίνκο, το περίμενα. Το αισθανόμουν πριν από την ψηφοφορία. Είναι απογοητευτικό. ένα από τα νέα στοιχεία αυτής της οδηγίας είναι ακριβώς αυτή η έννοια της ευθύνη Είναι ένα νέο ευρωπαϊκό μέσο, είναι η προστιθέμενη αξία αν θέλετε. Έτσι πίστευα εγώ, αλλά δυστυχώς η Επιτροπή μου δεν το δέχτηκε. Τέλος, να πω ότι θα... Μα αποσύρω μάλλον το όνομά μου, αλλά θα διαβάσω προσεκτικά το κείμενο, πρέπει πάντα να το κάνουμε αυτό. Και ελπίζω ότι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να είσαστε προσεκτικοί στα νέα στοιχεία, όχι μόνο στο 9 και το 12, αλλά όπου ακριβώς έχει υπάρξει προστιθέμενη αξία από την ΙΝΚΟ σε αυτήν την οδηγία. Ελπίζω ότι η δική σας επιτροπή θα είναι λίγο πιο ρεαλιστική και λίγο λιγότερο ιδεολογική όταν αξιολογήσει το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει στο μέλλον θα πρέπει να ακούμε αυτά που λένε οι επιθεωρήσεις εργασίας, θα πρέπει να σεβόμαστε την κοινωνική εταιρικότητα και ελπίζω εσείς σαν Επιτροπή να βοηθήσετε να δημιουργηθεί ένα σωστό νομικό πλαίσιο για τις αποσπάσεις με αξιοπρέπεια. Δεν τα καταφέραμε στην Επιτροπή, να τα καταφέρετε εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν για το άρθρο 3. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται η δυνατότητα σημαντικής ε, ε, δραστηριότητας ή περιορισμένου αριθμού. Θεωρείται ότι ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι καθοριστικά για, την, για το χαρακτηρισμό του νομότυπου ή του παράνομου χαρακτήρα της απόσπασης. Γιατί με κάτι τέτοιο θα οδηγηθούμε στην κατάσταση πολλές βελγικές ε, επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητες στη Γερμανία, Γαλλία ή κατοχώρες δεν θα μπορέσουν να κάνουν αποσπάσεις εξαιτίας ε, της έλλειψης της βασικής δραστηριότητας ε, στις χώρες αυτές. Επίση, θα είναι δύσκολο το θέμα και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα χρειαστεί και αυτές να απολύσουν τις αποσπασμένες ή να, να μην προβούν στην, στην απόσπαση. Γιατί τελικά θα έχουν προτεραιότητα οι εργαζόμενοι της χώρας υποδοχής. Σε μερικές ε, περιπτώσεις ε, ε, έχουμε τα σημεία της απόσπασης που είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει αυτά να εξετάσουμε πριν να λάβουμε υπόψη τον περιοριστικό χαρακτήρα των σημείων του άρθρου 3 για τη βασική κυρίως δραστηριότητα. Συμφωνώ με τις προτάσεις σας για την πρόσβαση στην ενημέρωση, όχι μόνο για τους όρους πρόσληψης, αλλά και για τους ε, τρόπους ή τα μέσα ελέγχου που θα ισχύουν για τους εργοδότες. Θα πρέπει βέβαια να ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να απαιτηθεί από τον εργαδότη, ιδιαίτερα όταν είναι αλλοδαπός. Ε, θα πρέπει η πρόσβαση να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα για όλους. Και τέλος, κάτι που αναφέρατε, κυρία εισηγήτρια, στην πολύ εμπεριστατωμένη σας παρουσίαση προηγουμένως, στην υποχρέωση εξασφάλισης στον αποσπασμένο εργαζόμενο των εξόδων ε, μεταφοράς, ε, διανυκτέρευσης, διαμονής και διατροφής καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασης. Γιατί η κεντρική οδηγία, η βασική οδηγία δεν προβλέπει τέτοια υποχρέωση, γι' αυτό και καταθέσαμε τη σχετική τροπολογία, γιατί θεωρούμε ότι έχει τέτοιο δικαίωμα ε, ο εργαζόμενος να... Αλλά συμφωνώ ότι σε ό,τι αφορά τα μέτρα την αποζημίωση των εσόδων μεταφοράς διαμονής και διατροφής αρμόδιο είναι το κράτος της προέλευσης, ενώ για τον καθορισμό της ελάχιστης αποζημίωσης αρμόδιο είναι το κράτος μέλος υποδοχής. Είμαι πρόθυμη πάντως για συμβαστικές λύσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε μια νομοθετική διάταξη που θα είναι αμοιβαία ικανοποιητική για όλους. Ο κύριος Κοζουόφσκι. Ο κύριος Κοζόφσκι. Θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ εν συντομία στο άρθρο 3. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ανέντιμες πρακτικές και τους ανέντιμους εργοδότες, αλλά θα πρέπει να τιμωρούμε τους έντιμους και ειλικρινείς εργοδότες και να τους απογορεύσουμε ουσιαστικά να αποσπάσουν εργαζόμενους. Γιατί δεν μπορεί η μη τήρηση κάποιων στοιχείων του άρθρου 3 να μας οδηγεί στο χαρακτηρισμό της παράτυπης ή της παράνομης απόσπασης. Γι' αυτό και κατέθεσε την τροπολογία 30, 90 ε, που αναφορά τα αποτελέσματα της μερικής στήρησης του άρθρου 3. Προτείνουμε λοιπόν το κράτος της προέλευσης αλλά και το κράτος της υποδοχής να συνεργαστούν στενά και να καθορίσουν κάποιες διατάξεις που με βάση τη Σύμβαση Ρώμη 1 θα βελτιώσουν την κατάσταση των αποσπασμένων εργαζομένων. Πιστεύω ότι αυτή είναι πολύ καλύτερη λύση από το να καθορίσουμε τις συνέπειες της μη τηρής κάποιων σημείων του άρθρου 3. Γι' αυτό και παραλαμβάνω κατέθεσα την τροπολογία 90 προκειμένου να βελτιωθεί το άρθρο αυτό. Κυρία Σρέντερ και μετά Τσαμπόρη. Κυρία Σρέντερ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για μια πρώτη σύνοψη των όσων έχουμε συζητήσει στον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων. Ε, από κοινού κάτσαμε και με υπομονή εξετάσαμε το πώς θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινέ γραμμές. Συμφωνώ με την θέση ότι χρειαζόμαστε σαφή νομοθεσία, μια νομοθεσία η οποία θα πρέπει να είναι ε, ξεκάθαρη δηλαδή σε ό,τι αφορά την παράγραφο για τις πληροφορίες, θα πρέπει να μιλάμε για τις πληροφορίες και επίσης η παράγραφος που θα αφορά τις ε, επιτετραμένους θα πρέπει να αφορά τους επιτετραμένους. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι σε ό,τι αφορά τα άρθρα. Είναι δύσκολη η διαπραγματευτική κατάσταση και για την εισηγήτρια, γιατί θα πρέπει να πείσει τους συναδέλφους ότι οι τροπολογίες τους θα πρέπει να απευθύνονται σε, άλλ, για σε άλλα άρθρα. Είναι σημαντικές λοιπόν οι εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί. Συμφωνώ με τον ε, Στίβεν Χιούς. Μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε, να ξεκινήσουμε με τα βασικά άρθρα, να θέσουμε κάποιες γραμμές και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Γραπτή η πρόταση του Στίβεν Χιούς, την οποία και υποστηρίζω. Επίσης, συμφωνώ με την άποψή σας ότι χρειαζόμαστε καλή νομοθεσία προκειμένου να κάνουμε καλές διαπραγματεύσεις με τον συνομοθέτη, να εξετάσουμε ενδεχόμενους συμβιβασμού που έχουν επιτευχθεί και εκεί, για να τους ε, υιοθετήσουμε ενδεχομένω. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ιδάλω δεν θα τα καταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και υπάρχουν πάρα πολλέ συνεδριάσει οι οποίε προβλέπονται. Αλλά χρειαζόμαστε και το χρόνο μας για καλή νομοθεσία. Επίσης, συμφωνώ με αυτά που είπε η συγγήτρια ότι χρειάζεται η βέλτιστη πληροφόρηση των εργαζομένων. Συμπληρώνω και για τους εργοδότες χρειάζεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Αμφιβάλλω, αμφιβάλλω για το κατά πόσον μία και μόνη στο σελίδα δεν θα καταφέρει αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποχρεούνται να βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις κάθε φορά και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο προσανατολισμού μας. Μια σημαντική, ένα σημαντικό μέσο μπορεί να είναι μια ιστοσελίδα, όντως, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν φτάνει μια ιστοσελίδα. Γι' αυτό λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Δεν πιστεύω, όπως είπε η συγγήτρια και όπως παρουσιάζει η συγγήτρια ότι οι κανόνες του κράτους προέλευσης θα πρέπει να ισχύουν σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την ε, φροντίδα. Γιατί σε ό,τι αφορά την ελάχιστο μισθό, για παράδειγμα, ορίζεται την αρχική οδηγία ότι θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες του κράτους ε, εργασίας θα πρέπει να τα τηρήσουμε όλα αυτά για να μην περάσει έτσι εμέσως μια αλλαγή της αρχικής οδηγίας μέσω της τροπολογιών μας δηλαδή. Πιστεύω ότι το άρθρο 9 θα πρέπει να είναι ανοιχτό. Προκειμένου να μπορούμε να προσαρμοστούμε στην εκάστοτε κατάσταση. Τα υπόλοιπα πολύ απλά δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν είναι ρεαλιστικά συμφωνώ στην παρούσα φάση ότι οι κλασικές νομικές μορφές στην Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η επικουρικότητα, η διαφάνεια, σύμφωνη. Αλλά μια κλειστή λίστα θεωρώ ότι είναι κάτι το τελείως ε, ανεδαφικό. Δεν είναι εκτελεστική αυτή η οδηγία εφαρμοστική, θα πρέπει να βρούμε μορφές ελέγχου. Ενδιαφέρον ήταν ότι η συγγήτρια είπε ότι η επιθεώρηση δεν θα πρέπει να είναι περιοριστική. Ναι, μα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν θέλουμε να είναι περιοριστική η επιθεώρηση, θα πρέπει να προβλέπονται και εναλλακτικέ λύσεις. Και συμφωνώ με την Άντια πρέπει να σας πω ότι στη Γερμανία είχαμε πάρα πολύ καλές εμπειρίες με την αποκοινού αλληλεγγύη ευθύνη. Και στη Γερμανία έχουμε πολλές μικρές εξωτερικές ε, ε εταιρείε και εγώ είμαι από την Ανατολική Γερμανία και να σας πω ότι περισσότερες από τις μισές ε, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών δεν είναι γερμανικού δικαίου. Και τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά μας τι γίνεται με την κοινού και αλλαγή ευθύνη. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι νομική σαφήνεια σε πολλές περιπτώσεις και είναι σαφές ότι θέλουμε να μπορέσει η Γερμανία να διατηρήσει αυτό το σύστημα το οποίο είναι πολύ αξιοθαύμαστο. Αυτό ήταν εν συντομία, με μεγάλη συντομία, ε, Αυτά ήταν τα βασικά σημεία που ήθελα να σας παρουσιάσω. Νομίζω ότι όσο Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να είναι καλύτερη, να είναι, καλή νομοθεσία στην οποία θα καταλήξουμε. Ίσως να χρειαστούμε και πιο πολύ χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει αρχικά. Ο κύριος Ζωρή και μετά για την Πάουδερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω. Οι συνάδελφοι με κάλυψαν σε πολλά από τα σημεία που σκόπευα να αναφέρω. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9, το όλο θέμα της ανοιχτή ή κλειστή λίστας. Επιτρέψτε μου να πω ότι σέβομαι την κυρία Τουρμέν και την δουλειά της, αλλά για το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ φοβάμαι ότι δεν θα συμφωνήσω μαζί της. Δεν ξέρω αν είναι ιδεολογική η συζήτηση που έλαβε χώρα στην ΙΜΚΟ, για τη συντελική ανάλυση η ΙΜΚΟ υποστήριξε τη διαμόρφωση μιας κλειστής λίστας και εγώ συμφωνώ. Έχουμε μακρά εμπειρία στον τομέα αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε διάφορα προστατευτικά μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις ε, έγινε απόπειρα να δυσκολευτεί πολύ η κατάσταση για άτομα τα οποία έρχονται από άλλη χώρα. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μία ενιαία ώρα, την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Μιλάμε για την ε, κινητικότητα, μιλάμε για την ενιαία αγορά, μιλάμε για την δημιουργία θέσεων εργασία, νέων θέσεων εργασία. είναι όλα πρακτικά αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε λοιπόν νομική αβεβαιότητα και να μην περιπλέκουμε τα πράγματα και να προκαλούμε νομική αβεβαιότητα πολύ απλά γιατί κάποιες χώρες ίσως για πολιτικούς λόγους, θέτουν αυθαίρετα νέες ε, συνθήκες, νέους κανόνες, νέους όρους. Περιπλέκοντας τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η κλειστή λίστα μας εγγυάται τη νομική βεβαιότητα που χρειαζόμαστε. Μιλάτε για την ενιαία αγορά και θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχουν ομοιόμορφοι κανόνες σε όλη την Ένωση. Εκ παραλίλου, ασφαλώ μπορεί να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο. Ε, κατά την οποία θα υπάρχουν τακτικοί έλεγχοι και τακτικές, ε, ε, τακτική εξέταση της λίστας. Άρα προτείνω ίσως κλειστές λίστες, αλλά κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να επιγίνεται ένας έλεγχος, ίσως με πράξεις κατά εξουσιοδότηση, για να καταγράφεται η κατάσταση σε κάθε μέρος και αν θεωρηθεί ότι χρειάζεται επέκταση της λίστας, συμφώνει να γίνει, αλλά να ισχύει για όλη την Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν πιο σκόπιμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ενιαία αγορά και για τη λογική που κρύβεται πίσω από την αγορά. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ και τώρα και μετά ο Όλε Κρίστινσεν. Ευχαριστώ, λέει κυρία Μπάουερ. Δύο σχόλια να κάνω. Καταρχά θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο γιατί εξέτασα τις τροπολογίες και παρακολούθησα και την όλη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Μου δίδεται η εντύπωση ότι κάποιοι από του συναδέλφου μας και μάλιστα μεγάλο τμήμα της Επιτροπής μας εξετάζουν την οδηγία για τους αποσπασμένους λες και μιλάμε για κάποιο είδους έγκλημα, για κάποια εγκληματική δραστηριότητα. Τέτοια προσέγγιση ακολουθούν. Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Δεν ε, ε, υιοθετούμε, δεν δημιουργούμε έτσι καλή νομοθεσία, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω για την παράγραφο 12 συγκεκριμένα. Για την παράγραφο 12. Κατά κάποιο τρόπο θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική παράγραφο της πρότασης. 50 σελίδες τροπολογίες έχουμε για την παράγραφο αυτή οι μισές εξ αυτών ζητούν διαγραφή όλη τη παραγράφου, μισή παραγράφου, τμήματων τη παραγράφου και οι υπόλοιπε τροπολογίε έχουν να κάνουν με περικοπή τη παραγράφου αυτή. Μιλάμε για την παράγραφο για την αποκοινού και αλληλέγγυα ευθύνη σε ό,τι αφορά του υπεργολάβου. Είναι μεγάλο το εύρο. Σύμφωνοι. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι συμμετείχαμε και στην κατάρτιση προηγούμενων νομοθετημάτων και γνωρίζουμε πόσο ακαθόδες είναι το ζήτημα αυτό. Κάποιες, αρχε... Κάποιες χώρες δεν έχουν την αρχή αυτή στην ε, χώρια νομική πραγματικότητά τους. Άρα, είτε μιλάμε για τις εταιρείε ε, που είναι υπεργολάβοι και όταν μιλάμε για την ε, ευθύνη τους, πέρα από το βασικό εργολάβο, αυτό θεωρώ ότι επηρεάζουν πολύ τι αρχέ που ανέφερα στην αρχή τη παρεμβασή μου. Ξέρω ότι είναι πολύ ακαθόδες το θέμα αυτό και προχαλεί μεγάλο διχασμό, αλλά πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή την κατάσταση, να κοιτάξουμε την θέση του βασικού εργολάβου, που δεν έχει δικαίωμα να εξετάσει, να ελέγξει τους μισθούς, τις ε, λογαριασμούς του εργολάβου θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι, μετριοπαθείς στον τομέα αυτό και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια λογική λύση στη τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Όλε Κρίστενσεν και μετά Φίλιπ Μπενιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση της. Έχω μία ανησυχία, όπως σε κάθε περίπτωση που τύφεται το θέμα ε, του νοτου ανατολής-δύσης, τύφεται ιδεολογικό ζήτημα. Μετά από τους τελευταίους ομιλητές, μου δόθηκε ακόμα πιο έντονα η εντύπωση αυτή. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο θίγει και πλήττει διάφορες χώρες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μην θέσουμε νέα εμπόδια στην ιστορική αγορά, αντιθέτως να φροντίσουμε ότι όλα θα διεξάγονται ομαλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε την οδηγία που αντιμετωπίζουμε στην προκειμένη περίπτωση. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία σκοπό έχει να προστατεύσει τους εργοδότες, τους εργαζομένους και θα εγγυάται στους εργοδότες ε, τη σωστή τους λειτουργία. Το θέμα δεν είναι να δοθεί καλύτερη πρόσβαση σε απαταιώνες στα κράτη-μέλη από όπου και να προέρχονται. Όχι όταν κανείς μεταμένει από μια χώρα σε μια άλλη, θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται με τους όρους και τις συνθήκες που επικρατούν στο κράτος το οποίο μεταβαίνει. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν θα καταλήξουμε σε καμία σημαντική λύση των προβλημάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό θα το καταφέρουμε. Θα καταφέρουμε να ρυθμίσουμε τις διατάξεις αυτές, όσο περιπλοκές και αν είναι. Όταν μιλάμε για αλληλέγγυα ευθύνη, όταν μιλάμε για κλειστές λίστες. Όταν μιλάμε για κλειστές λίστες, ουσιαστικά ποιους προσελκύουμε. Τους απαταιώνες, οι οποίοι θα ξέρουν πώς θα χειριστούν αυτές τις λίστες. Αντιθέτως, εμείς θα πρέπει να προάγουμε τις ε, έντιμες επιχειρήσεις που θα προωθήσουν τον, ε, τον σωστό ανταγωνισμό. Οι νέοι τομείς οι οποίοι θα ανακύψουν και ενδεχομένως θα προκαλέσουν και κοινωνικό ντάμπινγκ ε, στην Ένωση έχουν να κάνουν συχνά με τον τομέα των μεταφορών, των οδικών και των αεροπορικών μεταφορών κυρίως. Σε αυτού του τομείς λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Νομίζω ότι αν δεν μπορέσουμε να αποδείξουμε, να τεκμηριώσουμε ότι ε, πρόκειται για ε, αποσπασμένο εργαζόμενο, θα πρέπει να εντάσσεται κανείς στο σύστημα της χώρας υποδοχής. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή προσέγγιση και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σωστό, λογικό, εύλογο πλαίσιο για τους εργαζόμενους που εργάζονται στο εξωτερικό. Ιδάλλως, το πρόβλημα αυτό θα συνεχίσει να μας πλήττει. Ευχαριστώ. Ο Φιλ Μπένιον και μετά το Μασμάν. Ευχαριστώ. Θα περιοριστώ στα άρθρα 11 και 12. Και θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου για την προσέγγιση της εισηγήτριας. Νομίζω ότι με ένα τέτοιο θέμα χρειαζόμαστε την υποστήριξη και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι είναι προς συμφέρον μας να έχουμε μια δογματική και απόλυτη θέση προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Γιατί δεδομένου του νομικού πλαισίου που μας περιέγραψε η κυρία Μπάουερ, έχουμε καθήκον απέναντι στους αποσπασμένους εργαζόμενους να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση που θα βρίσκει σύμφωνα τα κρατημέλη. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο ή σωστό ή δίκαιο να ζητήσουμε από ορισμένα κρατημέλη να τροποποιήσουν άρδιν τους εργατικούς τους κώδικες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα της οδηγίας. Γι' αυτό και για το άρθρο 12 κατέθεσα κάποιες τροπολογίες προκειμένου να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ενστενιστούν την αρχή της ισολόκληρων και ελέγγες ευθύνης και να μην τους την υποβάλουμε υποχρεωτικά. Πιστεύω μόνο ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε κάποια εναλλακτικά μέτρα ή να ενισχύσουμε κάποια ισχύοντα. Θα πρέπει να έχουμε και εναλλακτική λύση. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε μία μόνο λύση. Και πιστεύω ότι στις διμερείς ε, συζητήσεις που θα έχουμε με τον Επίτροπο θα το καταφέρουμε. Και οι περισσότερες τροπολογίες μου, ειδικά για τα άρθρα 11 και 12, στόχο έχουν την ε, πρόταση κάποιων εναλλακτικών λύσεων ε, σε ό,τι αφορά την ε, ισολόκληρη και από ευθύνη. Ευελπιστώ ότι σε συνεργασία με την εισηγήτρια θα καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες ώστε να συγκεντρώσουμε ευρία υποστήριξη. Κάτι βέβαια που δεν είναι σίγουρο. Ίσως τελικά επικρατήσει διάσταση απόψε μεταξύ μας για τα θέματα αυτά. Αν κάτι τέτοιο γίνει, τι να κάνουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον και ό,τι έγινε και ό,τι γίνει ας γίνει. Τώρα, για τις εργασιακές συνθήκες ποιος ποιες θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Πιστεύω ότι οι εργασιακές συνθήκες θα πρέπει να αφορούν το κράτος μέρος στο οποίο ε, εκτελείται η εργασία. Αλλά και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί αν η εταιρική έδρα της ε, νομικής οντότητας βρίσκεται αλλού, τότε κάποια θέματα θα πρέπει να συνδυάζονται με τον, το κράτος της έδρας. Θα πρέπει να δούμε ποιες εργασιακές συνθήκες ποια χώρα θα ισχύουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει, διαφαίνεται η πιθανότητα συμφωνίας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ήδη να ανασκουμπωνόμαστε για πόλεμο από τώρα. Ο Τόμας Μαν και μετά η Ρίτα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Όλε Κρίστενσεν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κίνδυνος που προκύπτει είναι ότι μπορεί τελικά να πλεχτούμε σε μια συζήτηση τεχνητή. Μεγάλες, μικρές χώρες, ε, ε, βορράς κατά του νότου. Αυτό δεν είναι σωστό και δεν έχει νόημα. Το θέμα δεν είναι αυτό μάλλον. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά υπό τις σωστές συνθήκες. Οι, Γερμανές, ε, Γερμανοί λένε ότι, μάλλον ακούγεται ότι οι Γερμανοί θέλουν κάτι να αποφύγουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να ξέρουμε αν πρόκειται για νόμιμα εργαζόμενους ή για λαθρέα εργαζόμενους. Το θέμα είναι να έχουν τα σωστά ε, πιστοποιητικά, τα σωστά έγγραφα. Γι' αυτό θα πρέπει να καταλαβαίνουν τη γλώσσα τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζητάμε μεταφραστές αλλά αυτό ίσω να κοστίζει πολύ, ίσω να διαρκεί υπερβολικά πολύ χρόνο. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί λοιπόν. Χρειαζόμαστε κανόνε όπου θα ορίζεται και θα καθορίζει η αρχή της ε, χώρας ε, προέλευσης. Οι επιχειρήσεις ε, οι οποίες θέλουν να καταχραστούν την κατάσταση και στη δική μου χώρα υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, δεν είναι όλες καλές και οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν τις πιο φθηνές υπηρεσίες από όπου και αν έρχονται το θέμα λοιπόν δεν είναι θέμα Ανατολής ε, κατά της Αντιθέτως, αναφέρεται ότι θέλετε μια κλειστή λίστα. Αυτό θα το έχει δίκαιο θα το καταχραστούν οι απαταιώνες. Αυτό δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Οι ανοιχτές λίστες, Νάντια, δεν έχουν ως σκοπό να μπορούν να πούν ε, τα κρατημέλη και οι επιχειρήσεις ότι θέλουμε να τις υπονομεύσουμε. Αντιθέτως, αν ε, προκύψουν σε καταστάσεις θα πρέπει να προσθεθούν στην λίστα. Αυτό δεν μπορεί να ε, εμπλέξει κλειστές λίστες γιατί αυτό θα το καταχραστούν πολύ. Παντού υπάρχουν σωστοί και καλοί εργαζο... εργαζόμενοι και εργοδότες που φροντίζουν να πληρώνουν τις εισφορές τους στα Ανατολή και Δύση και αυτούς θα θέλουμε να προωθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ιστορική Αγορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό θεωρώ. Συμφωνώ και με την ε, κυρία Σρέντερ που μίλησε για τους κανόνες της ε, χώρας προέλευσης που θα πρέπει να ισχύουν. Και εδώ χρειαζόμαστε σωστή πληροφόρηση όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες να ξέρουν τι τους αφορά γιατί πολλοί μου λένε ότι δεν ξέρουν οι εργοδότες τι χρειάζεται να κάνουν. Μα δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να ξέρουν τι ισχύει. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και για εργοδότες και για εργαζόμενους. Το κατά πόσο αυτά μπορούν να, να επιτευχθούν με μία σελίδα, δεν νομίζω. Και σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ιδεολογικό αγώνα. Θα πρέπει. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις νόημες δραστηριότητε. Και αυτό, για να το πετύχουμε, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος τους κανόνες που ισχύουν. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Τελευταία παρατηρήση στις οικοδομές. Ένα μόνο παράδειγμα αναφέρω. Στη Γερμανία, στις οικοδομές, έχουμε μεγάλο έλεγχο επειδή θέλουμε να ξέρουμε το ύψος της μαύρης εργασίας. 660 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει κάθε χρόνο η παράνομη εργασία. Μα καταλαβαίνετε το ύψος του προβλήματος, ανεξάρτητα από το που έρχονται οι εργοδότες, αν πληρώνονται σωστά, αν έχουν τις διακοπές τους, αν έχουν όλα τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να έχουν, όχι μόνο για να χτίζουν ε, τύχη, στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα αυτό, αλλά για να έχουμε διαφάνεια. Αυτή τη διαφάνεια θα πρέπει να επιδιώξουμε. Θα ήθελα στις συζητήσει μας, στις μελλοντικέ να υπάρχει και μια, ένα κοινό πνεύμα για να αναπτύξουμε κοινέ γραμμές, για να μην ξαναπέσουμε στις παλαιές διαμάχες, στις παλιές διαφωνίες. Γιατί δεν αξίζει. Χρειαζόμαστε καλή, ακριβή νομοθεσία, κοινή νομοθεσία. Γιατί πιστεύω στο καλό του που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, αλλά και στο καλό που υπάρχει εδώ στην Επιτροπή. Απλά να ακούμε ένα τον άλλον. Είμαι βέβαιος ότι στην περίπτωση αυτή θα πετύχουμε ένα καλό ορόσημο στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, κυρία Όμεν Ρόιτεν, και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ξαναρώτησα πριν από λίγο. Το 2006 καταρτήσαμε μία έκθεση για την οδηγία για τους αποσπασμένους και ήταν η κυρία Σρόντερ η συγγήτρια και θυμάμαι ότι και εγώ ήμουν συντονίστρια και μαζί με τον Στίβεν κάναμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ε, τότε διαπιστώσαμε, Πρόεδρε, ότι η απόσπαση ε, είναι υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας και ότι είναι θετικό ε, θέμα αλλά ότι υπήρχαν και πολλά, ε, πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την απόσπαση και τα οποία προβλήματα προσπαθήσαμε να τα επιλύσουμε τότε. Και ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε πέρα από κάθε προστατευτισμό και να αποφύγουμε τη δημιουργία παρεξηγήσεων. Αυτό το είχαμε διαπιστώσει από τότε. Και τώρα είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό αυτό ελεύθερη κυκλοφορία, καλές ε, θέσεις εργασίας, αλλά αποφυγή παρεξηγήσεων. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ κάποιων στοιχείων και τα άρθρα τα οποία αναφέρθηκαν είναι όντως πολύ σημαντικά. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη καταχρήσεων, θα πρέπει να υποβάλουμε τα σωστά κριτήρια. Μια πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει κλειστή λίστα ή ανοιχτή λίστα η κλειστή λίστα έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά η ανοιχτή λίστα ταιριάζει πιο πολύ στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρώ ότι η ανοιχτή λίστα δεν θα πρέπει να τύχει κατάχρηση. Γι' αυτό λοιπόν οι κανόνες θα πρέπει να είναι όχι μόνο ξεκάθαροι, αλλά αν κάποια χώρα θέλει να έχει επιπλέον κανόνες λόγω της λίστας, θα πρέπει εκ των προτέρων να ορίζει η χώρα εκείνη να ορίζει και να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους κανόνες αυτούς προκειμένου να τις ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία, Πρόεδρε, ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ενός συμβιβασμού. Αυτό αφενός. Κατά δεύτερον, και τότε το είχαμε εξετάσει, είχαμε μιλήσει για τους αυταπασχολούμενους. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και νομίζω ότι και στον τομέα αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και προς αυτήν την κατεύθυνση κατεύθυνση τροπολογίες και σε διαφορά την παροχή πληροφοριών. Θεωρώ ότι μπορούμε πολλά να πετύχουμε. Πολύ περιθώριο βελτίωση υπάρχει για τον ρόλο της επιθεώρησης. Θεωρώ ότι είναι κάπως αδύναμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσουμε λοιπόν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιθεωρήσεις για την αλληλεγγύη. Εδώ έχω κάποια σημεία να ασκήσω κριτική. Ε, συνάδελφοι Μπελέτ και Μπροκ και εγώ συνυπογράψαμε κάποια σχόλια τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να τα συμπεριλάβει η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή. Θετικά λοιπόν τα σχόλια μου, όχι μόνο επειδή είναι φίλη μου η Τανούτα, αλλά επειδή θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε καλούς συμβιβασμού, Αρκεί να πείσουμε ότι δεν είναι ο σκοπός μας ο προστατευτισμός. Όχι. Σκοπός μας είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και θεωρώ ότι η Ντονούτα συμφωνεί σε αυτό. Θα περιμένω λοιπόν τη διαμόρφωση συμβιβασμών, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Οι συμβιβασμοί θα εξαρτηθούν από την καλή θέληση όλων σας. Έχετε δίκιο που επιμένετε στο συγκεκριμένο. Θα επανέλθω τώρα σε τρεις πλευρές. Καταρχάς, σε σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Ομενρόιτεν με τις επιθεωρήσεις. Και εδώ έχουμε καταθέσει κάποιες βασικές τροπολογίες για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις ελεγκτικές υπηρεσίες, ανάμεσα στις επιθεωρήσεις ιδιαίτερα στον τομέα των εργοταξίων της οικοδομής, ξέρετε πόσο διαφέρουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα και καμία τελικά χώρα, καμία υπηρεσία κοινοτική συγγνώμη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να ανασυνθέσει αυτό το πάζολ των εθνικών νομοθεσιών και δυστυχώς αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των σύγχρονων δουλεμπόρων, αυτών των δουλεμπόρων ενοικίασης καταλημάτων απαράδεκτων. Σχετικά με τον συντονισμό πάντα λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποια πρόοδος. Για τον κατάλογο. Εδώ κατανοώ και συντονίζομαι με την κυρία Σρέντερ. Κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουν πόλεμοι καινούργοι και ιδεολογικές διαφωνίες. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία μας καθοδηγεί συστηματικά. Είμαστε στην υπηρεσία της βελτίωσης της κατάστασης των εργαζομένων. Και βασική αρχή λειτουργίας μας είναι ότι σε ισότητα απασχόλησης αντιστοιχεί ισότητα δικαιωμάτων. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο φανταζόμαστε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει επιτόπου. Και ο στόχος της διαπραγμάτευσης είναι να εγγράψουμε αυτή τη βασική αρχή στις περιοχές όπου εργάζονται ε, οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με μία άλλη αρχή θα έλεγα βασική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ στον κοινωνικό τομέα δεν είχε θα έλεγα ένα επίπεδο θα έλεγα εφαρμογής των κανόνων της ιδιαίτερα μεγάλο. Η αποδοχή των κοινοτικών κανόνων δηλαδή ήταν περιορισμένη. Υπήρξε όμως μια βασική αρχή η οποία έγινε πάντα δεκτή. Ήταν η αρχή της μη υπαναχώρησης. Πέραν αυτού λοιπόν και εφόσον εμένουμε σε έναν κλειστό κατάλογο στον τομέα της δυνατότητας των εθνικών επιθεωρήσεων, σε αυτή την περίπτωση θα παραβιάσουμε την αρχή της συνθήκης σχετικά με την αρχή της μη επαναχώρησης στον κοινωνικό τομέα. Και η τρίτη σειρά των επιχειρημάτων αφορά προφανώς το άρθρο 12 Εγώ δεν έχω εντυπωσιαστεί από τις ε, τροπολογίες διαγραφής που έχουν κατατεθεί. Ξέρω ότι στην ουσία σε πολλές εκθέσεις καταντίθενται προτάσεις διαγραφής κάθε παραγράφου και στο τέλος καταλήγουμε σε καλές συμβιβαστικές προτάσεις. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και νομίζω ότι η Εντίθ το είπε αλλά δεν είναι μαζί μας τώρα ότι δεν θα πρέπει εμείς να θεωρούμε εκ των προτέρων την διαδικασία της απόσπασης σαν μια ύποπτη διαδικασία. Κοιτάξτε όμως κάποιες ε, αγορές εργασίας όπου η σύγχυση ανάμεσα στους αποσπασμένους εργαζομένους και τους εργαζομένους στη μαύρη αγορά είναι σαφής. Υπάρχει θα έλεγα μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων είναι ελάχιστα. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει ο κατάλογος αυτός να διευρυνθεί. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντυπήσει σωστά το θέμα του προβλήματος στον τομέα των οικοδομών. Αλλά γιατί όχι η Γεωργία γιατί όχι επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, μιλάμε για μια καταστροφή. Οι ύποπτες δραστηριότητες πολλαπλασιάζονται με φρικτό και απαράδεκτο τρόπο. Και στις μεταφορές επίσης, και στις μεταφορές. Ελπίζω λοιπόν αντίθετα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με διάφορους τρόπους, θα δούμε πώς, για να διευρύνουμε τον κατάλογο αυτό επί του, οποίου, επί του οποίου θα βασιστούμε για να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Έχετε τον λόγο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε χρόνο πια. Αφού μίλησα, ζητώ συγγνώμη που θα το κάνω. Όχι πάνω από τέσσερα λεπτά. Σε δύο λεπτά. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλες αυτές τις 800 τόσες τροπολογίες. Καταρχάς, θα πρέπει να μιλήσουμε για ξεκάθαρους και ε, εύληπτους κανόνες. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ. Το μέσο είναι η επιβολή της οδηγίας και όχι η αλλαγή στη βασική οδηγία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, διότι στην αρχική οδηγία σχετικά με την επιστροφή της κατοικίας και της τροφής υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη φράση. Ενώ κάποιες τροπολογίες αλλάζουν, αλλοιώνουν θα έλεγα το άρθρο αυτό. Αυτό εξηγεί γιατί η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για τα καταλήματα των ε, εργαζομένων αντικατοπτρίζεται με προσεκτικό τρόπο στα άρθρα 3 και 11.5. Δεν πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε σε βάθος τη βασική οδηγία 96-71 γιατί πράγματι de facto το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις χωρίς να αλλάξουμε τη βασική οδηγία. Ένα δεύτερο σχόλιο. Σε ορισμένες από τις τροπολογίες γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα άρθρα της αρχικής οδηγίας, στα 3, στα 4, στα 5 αναφέρονται πάρα πολύ συχνά. Το πρόβλημα με την αρχική οδηγία είναι ότι τα άρθρα 4 και 5 σαν παράδειγμα ορίζουν με πολύ γενικό τρόπο τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Προσπαθούμε εμείς να αναλύσουμε με πιο προσεκτικό τρόπο στην οδηγία επιβολής. Αν τώρα ξεκινάμε από τις αρχικές διευκρινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε απλά να σεβόμαστε τη γενική διατύπωση της αρχικής οδηγίας, τότε φοβντάζομαι ότι θα καταλήξουμε σε αντιφατικά αποτελέσματα και μη αναμενόμενα. Υπάρχουν επίσης ορισμένες τροπολογίες σε συγκεκριμένα άρθρα που συγκεντρώνονται στην δυνατότητα οικονομικής στήριξης. Εμείς στην αρχική μας πρόταση προσπαθήσαμε στο άρθρο 8 να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Αν προσπαθήσετε και εσείς στα πλαίσια των συμβιβαστικών τροπολογιών γύρω από την αλλαγή του άρθρου 8, μετά από μακρές συζητήσεις νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι είναι σαφείς οι λόγοι για την αλλαγή του 8. Τώρα σχετικά με την διάκριση ανάμεσα στο 9 και 10. Νομίζω ότι η συγγήτρια είπε ήδη ότι υπάρχει διαφορά. Το 9 είναι τα εθνικά ελεγκτικά μέτρα, ενώ το 10 είναι οι επιθεωρήσεις οι κοινοτικές. Πέραν αυτών λοιπόν, μετά από τις συζητήσεις που έγιναν και, και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, ίσως κάποια στοιχεία καινοτόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έχουν την πρόθεση να μειώσουν τις, επι, τις ελεγκτικές δυνατότητες, και να αλλοιώσουν την αρχική πρόταση. Η αρχική πρόταση έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται επιπλέον θέματα να τίθενται στους παροχείς υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και σχετικά με τα πιστοποιητικά σαν παράδειγμα τα οποία θα πρέπει να εκδίδονται για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εργάζονται στα πλαίσια περιβάλλοντος χρήσης αμοιάντου κτλ. Αυτές είναι ρυθμίσεις που αφορούν το άρθρο 9 και δεν θέλουμε εμείς να αλλάξει η αρχική πρόταση, δεν θέλουμε να ανοίξουμε νέες δυνατότητες στην αγορά και οι πιο αντιφατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα δύσκολα άρθρα έχουν εντοπιστεί, οι συζητήσεις ήταν δύσκολες, όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε όμως την οδηγία αυτή και έναν καλύτερο και μεγαλύτερο σεβασμό των δικαιωμάτων των αποσπόμενων εργαζομένων και όχι ένα κείμενο το οποίο δεν θα είναι σε θέση να εφαρμοστεί. Σκοπεύω λοιπόν να συνεργαστώ επικοδομητικά με το Κοινοβούλιο και να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες σε αυτά τα δύο άρθρα, τα οποία επαναλαμβάνω δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ήταν πάντα και όταν κάναμε την αρχική πρόταση και το γνωρίζαμε. Σας ευχαριστώ. Η συγκήτρια τώρα. Ήταν όντω εκτενέστατη συζήτηση, αλλά δεν μπορώ να σα δώσω παρά μόνο πέντε λεπτά για σήμερα για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είναι και πολύ εύκολη αυτή η, η οδηγία και αυτή η υποχρέωση. Σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση του κυρίου Χιούς να την ε, αντιστροφή ε, της μεθοδολογίας ε, και την αντιστροφή των σημείων που θα επεξεργαστούμε, αλλά ήδη ξεκινήσαμε με την επεξεργασία των άρθρων. Θα έλεγα λοιπόν να μην αλλάξουμε αυτή τη σειρά, να συνεχίσουμε έτσι όπως ξεκινήσουμε, γιατί αν απομακρυνθούμε τώρα από αυτή τη σειρά θα δημιουργηθεί ένα χάος και μια σύγχυση. Σας ευχαριστώ κύριε Χιούς ε, για την πρόταση και τα άρθρα 9, 3, 9, 11, 12 είναι δύσκολα άρθρα, επίμαχα, θα χρειαστούν μακροχρόνια συζήτηση. Θα ασχοληθώ το συντομότερο δυνατό με τις, ε, συμβεστικούς, ε, με, τους, με τις συμβεστικές τροπολογίες ώστε να έχουμε μια βάση για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και κυρίως ε, σε αυτά τα άρθρα επικεντρώνομαι. Σε ό,τι αφορά την Άντια Χίρς, ήθελα να σου πω, Νάντια, ότι γενικώ όταν ε, μιλώ με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, μου λένε ότι οι διατάξεις ε, της Γερμανίας είναι καλές γιατί είναι διαφανείς. Γνωρίζει ο καθένας από την αρχή ε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες διαφανείς ε, ευανάγνωσες διατάξεις και είναι πολύ πιο εύκολο και για τον εργοδότη να, το, να καταλάβει τις υποχρεώσεις του και να προετοιμαστεί γι' αυτό. Γι' αυτό όλοι είναι ικανοποιημένοι με τις γερμανικές διατάξεις. Και αν ε, υποβάλουμε τέτοιες ε, διατάξεις, αυτή την οδηγία, ώστε να είναι διαφανείς, ευανάγνωστες, αντικειμενικές, να γνωρίζει από την αρχή ο καθένας τι τον περιμένει και πώς θα πρέπει να προετοιμαστεί, σίγουρα θα περιορίσουμε και τον αριθμό των ε, ανέντιμων ε, επιχειρηματιών γιατί θα τους δυσκολέψουμε ε, τη δυνατότητα καταχρήσεων. Ευχαριστώ και την Έμιλη που με ενημέρωσε για τις συζητήσεις στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Θα συζητήσουμε τις προτάσεις σου και θα δούμε με ποιο τρόπο θα Διαθετήσουμε μερικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά την κυρία Σξιντλεύσκα. συμφωνώ ότι το γεγονός που χαρακτηρίζει την απόσπαση, δηλαδή σημαντική ε, δραστηριότητα, η μεγαλύτερη δραστηριότητα στο, στη χώρα προέλευσης είναι όντως επίμαχο σημείο, γιατί ακόμη και για μεγάλες επιχειρήσεις ε, είναι δύσκολο να το υλοποιήσουμε και μερικές φορές αποκλείεται ο χαρακτηρισμός της, πραγμα... απόσπασης, παρόλο που θα πρόκειται για πραγματική απόσπαση εξαιτία του κριτήριου αυτού. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν. Ελίζαμπεθ, εγώ ουδέποτε δεν είπα ότι θέλω να περιορίσω ε, τις επιθεωρήσεις ή να τις καταστήσω πιο περιοριστικές. Το αντίθετο. Εγώ είμαι υπέρ της εξάλληψης των ανέντιμων επιχειρηματιών, της πάταξης της ανέντιμης συμπεριφορά και δεν είπα ότι θέλω να είναι πιο ε, περιοριστικές οι ε, επιθεωρήσεις. Δεν είπα θέλω να τις περιορίσω, θέλω η ε, έλεγχη να είναι σαφής και διαφανής. Γιατί σίγουρα όσο περιοριστικής και αν επιθεωρήσεις, αν είναι ε, ε, ανέντιμος ο επιχειρηματίας, ο εργοδότης, θα φροντίσει να τις παραγκάψει ούτως ή άλλως. Σε ό,τι αφορά τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Σόγκορ, σίγουρα με την οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Μας ενδιαφέρει η ενιαία αγορά. Και όλε Κρίστενσεν, θα ήθελα να πω ότι εγώ εκτιμώ απεριόριστα την αρχή της αλληλεγγύης. Και παρόλο που ακούω πολλές ε, ε, απόψεις για τους αποσπασμένους εργαζόμενους είτε από την Ανατολική είτε από τη Δυτική Ευρώπη. Εγώ είμαι Ευρωπαία παρόλα αυτά και προσπαθώ να συμβάλλω ε, στη διαμόρφωση ενός δικαίου που θα εξυπηρετεί και τις 27 χώρες, που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και ισότιμους κανόνες για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει εδώ καμία ιδεολογική προσέγγιση εκ μέρους μου και καμία μεροληψία. Είπε και ο Τόμας Μαν ότι παντού, σε όλες τις χώρες έχουμε και καλούς και κακούς εργοδότες. Σε όλες τις χώρες έχουμε και έντιμους και ανέντιμους εργοδότες. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου έχουμε ε, δύο είδη εργοδοτών. Αυτόν ε, τον εργοδότη που αποσπά του εργαζόμενους και του εργοδότη που τις λαμβάνει. Και οι δύο εργοδότε θα πρέπει να γνωρίζουν τι ε, ελέγχου θα υποστούν και τι πληροφορίες θα πρέπει να δώσουν και τι πρόσβαση θα του εξασφαλιστεί και τι ενημέρωση οφείλουν να κάνουν. κύριε Μπένιον, Παρακαλώ ολοκληρώστε κύριε εισηγήτρια, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών και τις διαφορετικές τους προδιαγραφές. Θα πρέπει να δώσουμε διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη να, να διαλέξουν το μέσο που θα εξασφαλίζει αυτή την αρχή της αλληλεγγύης και την αλληλέγγυη ευθύνη. Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε καλές νομοθετικές διατάξεις που θα είναι ευανάγνωστες, αποτελεσματικές, διαφανείς. Και μάλιστα έχω και μια πολύ καλή πρόταση του Τόμας Μαν εδώ. Πρότεινε ο κύριος Μαν να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση και να αποφύγουμε τα παλιά στερεότυπα και τις παλιές συγκρούσεις. Μακάρι ήθε είμαι διαλλακτική, ανοιχτή, πρόθυμη και θα δείξω κατανόηση και στις προθέσεις σας και στις προτάσεις σας. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς αυτό και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της και πολύ σωστή πρόταση για να διευκρινιστούν ορισμένα άρθρα. Είμαι ανοιχτή λοιπόν σε περαιτέρω συναντήσεις για να διαλευκάνουμε όλα αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ. Ε, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Λοιπόν, η νομική επιτροπή θα ψηφίσει στις 19 Μαρτίου. Συνεπώς εμείς θα κληθούμε να εξετάσουμε στις 20 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε την επομένη. Αυτά. Τελειώσαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Το τελευταίο θέμα για σήμερα... Το 39 η έκθεση της Επιτροπής μας για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ουγγουρεάνου. Very brief. As a draft person, uh, I... Είμαι πολύ σύντομος. Από πλευράς της Επιτροπής Απασχόλησης, η γνωμοδότηση θα εξετάσει τα εξή σημεία. Καταρχάς, ε, την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός ε, μεταξύ της Επιτροπής της ε, Πολιτικής Απασχόλησης και των στόχων του 2020, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε τις βασικούς πυρήνε, τι βασικέ πηγέ θέσεων απασχόληση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα βασικά οικονομικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί έχουν να κάνουν με τομεί που αφορούν τις επιχειρήσεις και αυτό ασφαλώς επηρεάζει το ποσοστό απασχόληση σε όλες τις χώρες. Άρα από την πλευρά αυτή το άρθρο 2 της γνωμοδότησης αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τα SGEIs από πλευρά της απασχόλησης. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, ιδιωτικοποίηση μη παραγωγικών επιχειρήσεων. Τελευταίο, τέταρτον και τελευταίο, πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια εξαίρεση από τους κανόνες για την κρατική βοήθεια προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές γιατί αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση των θέσεων εργασία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ο κ. Σέρκας και μετά αυτοί όλοι οι ομιλητέ. Ο κ. Σέρκας. Ευχαριστώ. Θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την πορεία των εργασιών ε, επί της έκθεσης αυτής. Μας ενδιαφέρει πολύ η πολιτική ανταγωνισμού και νομίζω ότι η υποχρέωση της Επιτροπής μας είναι να θετήσουμε διαφορετική προοπτική, διαφορετικό πρίσμα. Όλες οι προοπτικές είναι ε, εύλογες, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το δικό μας πρίσμα, δηλαδή σε ποιο βαθμό η πολιτική ανταγωνισμού συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ε, εργασίας και να δούμε μήπως ε, όχι μόνο την αναβαθμίζει αλλά την υποβαθμίζει σε μερικές περιπτώσεις. Οπότε, όπως είπε ο κύριος Ογκουράν, θα πρέπει να δούμε πώ μερικέ φορέ η πολιτική ανταγωνισμού έρχεται αντιμέτωπη στι κοινοφελεί υπηρεσίε. Δεν μπορεί και οι κοινοφελεί υπηρεσίε να υπόκεινται στι επιταγέ τη πολιτική ανταγωνισμού. Θα υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίε. Αν θέλουμε οι κοινοφελεί υπηρεσίε και αυτέ να υπόκεινται στην πολιτική ανταγωνισμού, είναι σαν να στερούμε σε ορισμένου ανθρώπου την πρόσβαση σε αυτές τις κοινοφιλείς υπηρεσίες. Γιατί σίγουρα δεν θα είναι οι κανόνε αγοράς που θα ενδιαφερθούν να εξασφαλίσουν κοινοφιλείς υπηρεσίες στους άπορους ε, ή σε αυτούς που περισσότερο τις χρειάζονται. Άλλωστε, αυτό λέει η συνθήκη και τα παραρτήματά της. Θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε λοιπόν την έκθεση αυτή προσθέτοντας το πρίσμα το κοινωνικό και το πρίσμα της απασχόλησης στα θέματα της πολιτικής ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι θα είναι πρόθυμος για περαιτέρω συζήτηση ο εισηγητή μα. Τώρα, δεδομένου του προχωρημένου τη ώρα, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε σήμερα τη συζήτηση και να προβλέψουμε προθεσμία για τι τροπολογίε. 27 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Η εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών θα λάβει χώρα στις 20 Μαρτίου και η ψηφοφορία στις 20 Μαρτίου. Η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή θα ψηφίσει στις 21 Μαρτίου τη δική της έκθεση. Επειδή ακριβώς ε, είναι πολύ βραχύβιες οι προθεσμίες, παρακαλώ τις τροπολογίες στα αγγλικά για τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, σας εύχομαι καλό απόγευμα και σας δίνω ραντεβού για την προσεχή μας συνεδρίαση το μήνα Μάρτιο. Καλό σας μεσημέρι.